Okay, ladies and gentlemen, if I can reconvene the meeting. We have uh, this... Έχουμε λοιπόν σήμερα το πρωί ακόμα μερικά, μερικούς από τους συντονιστές των ΔΕΔ και μετά θα έχουμε και τον Επίτροπο, τον Αντιπρόεδρο κύριο Κάλας και ε, όλα αυτά μέσα στο χρόνο που γνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένος. Επομένως το σφυρί μου θα λάμψει δια της παρουσίας του και δια του ήχου του. Θα πρέπει λοιπόν ε, να μην μαλώνετε μεταξύ σας όπως έγινε κάποια άλλη στιγμή, αλλά θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσετε το χρόνο σας έτσι ώστε ε, να θέτετε ερωτήσεις εις τους συντονιστές. Και επίσης και με όλο σεβασμό προς τους συντονιστές ε, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας, ε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως τα θέλουμε και επομένως 10 ε, λεπτά και για τους συντονιστές, 2 λεπτά για τους ερωτώντες από την Επιτροπή. Βοηθήστε με λοιπόν και η κυρία Τικάου όταν στις 11 θα πάρει τη θέση μου, βοηθήστε την και εκείνη. Θα είμαστε και οι δύο εξαιρετικά ευγνώμονες. Ξεκινούμε λοιπόν με τον επόμενο συντονιστή. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα προτεραιότητας 1 που είναι ο σιδηροδρομικός, γραμ... Ε, σιδηροδρομικός άξονας Βερολίνο, Βερόνα, Μιλάνο, Μπολόνια, Νάπολη, Μεσίνα, Παλέρμο. Ο εισηγητής, ε, συντονιστής μάλλον ο κύριος Πατκόξ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι πάλι εδώ στο Κοινοβούλιο. Τον Ιούνιο του 10 ε, πήρα την ε, θέση αυτή ε, και μετά από 7 μήνες κάναμε την πρώτη ενδιάμεση αξιολόγηση. Εν τω μεταξύ έχουν λάβει χώρα 19 αποστολές και θεωρούμε ότι από την τελευταία έκθεσή μας πολλές πρόοδοι έχουν γίνει. Να σας πω τώρα γρήγορα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Για τους πρώτους μήνες της περίοδου που ανέλαβα συντονιστής, ε, είχα κάποιες προτεραιότητες, ε, δηλαδή τον υπολογισμό του κόστους για το τούνελ στο Πρένερο και βεβαίως να λύσω προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή της Ιταλίας και της Αυστρίας τα κονδύλια ήταν ε, ε, αρκετά, αλλά παρόλα αυτά έλειπαν ε, αρκετά εκατομμύρια ευρώ που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν μέχρι το 2013 και όμως δεν είχαν αρχίσει στην ουσία να εκταμιεύονται και επομένως έπρεπε να γίνουν κάποιες διευθετήσεις και να γίνουν έλεγχοι πολλαπλής συμμόρφωσης και ρεσιμότητας. Έπρεπε επομένω να γίνουν και κάποιε αξιολογίε σχετικά με το συνολικό φάκελο, το πόσο, το πόσο δηλαδή θα κόστιζε στο σύνολο ε, το ε, έργο ε, αυτό. Επίσης έπρεπε να έχουμε τις επίσημες, την επίσημη μάλλον αδειοδότηση από τα κράτη-μέλη για να ξεκινήσουν τα έργα ε, και βεβαίως και συνεργασία και τις σχετικές αδειοδοτήσεις από τους σιδηροδρόμους της Αυστρίας και της Ιταλίας, τελικώς δε ε, και το μερίδιο της εθνικής χρηματοδότησης. Όλες αυτές οι προτεραιότητες και όλες αυτές οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν και στο Innsbruck πριν από λίγο καιρό ξεκινήσαμε τη φάση 3 και άρα τώρα μπαίνουμε στην κανονική ε, δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαδικασία ήταν πραγματικά ε, ουσιοδέστατη για την ε, ολοκλήρωση του έργου. Από εδώ και πέρα ξεκινήσαμε την οδό χωρίς επιστροφή. Ε, οι Υπουργοί όλοι και Μάστερ, καθώς επίσης και ο Επίτροπος ε, Κάλλας, ε, συναντήθηκαν για να λύσουν και τελικά προβλήματα, καθώς επίσης και η ανάδοχος τεχνική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την διόρυξη του τούνελ και αυτή έχει συνεργαστεί μαζί τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι συνεισέφεραν εις την προσπάθεια αυτή και επομένως εγώ δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα άτομα. Ενδεχομένως ο κύριος Μπουργμάιστερ της BBT ε, δούλεψε περισσότερο έτσι ώστε να εκπονήσει το master plan επί του οποίου συμφώνησαν όλοι. Μέχρι το 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και το τούνελ αυτό. Όσον αφορά την ε, υποδομή, ε, είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής ταυτόχρονα και στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της σιδηρογραμμής. Στην Αυστρία τώρα, στο βόρειο τμήμα, ε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί 41 χιλιόμετρα με, πολλές, με πολλά τούνελ, σύραγγες ε, και πολλή τεχνική δουλειά. Έχουν, ε, έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει τα έργα πολιτικού μηχανικού και ε, πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έκανα πολλές επισκέψεις εκεί και τα έργα μηχανικού που έχουν γίνει εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όσον αφορά το γερμανικό κομμάτι νότια του ε, Μονίχου, μέχρι τώρα μονάχα υπάρχει ε, ο σχεδιασμός επιχάρτου το σχέδιο, ε, το, σχέδιο εφαρμογής ε, που είχε εκπονηθεί πέρσι έχει καταλήξει ότι το κόστος θα είναι 2,6 ε, εκατομμύρια τα οποία έχουν ενταχθεί στην αναλυτική διαδικασία. Γίνεται προσπάθεια προόδου και στο κομμάτι αυτό και στο 13 Ιανουαρίου στο Ρόσενχάιμε θα γίνει μια συνάντηση ε, σε επίπεδο υπουργών ε, ε, ο υποφαινόμενος ως συντονιστής, ο Γερμανός υπουργός και ο Αυστριακός υπουργός, έτσι ώστε να υπάρξει υπουργική απόφαση για να προχωρήσουμε. Βεβαίως είναι πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά ε, πρόκειται για ένα βήμα απαραίτητο έτσι ώστε να μπουν στη διαδικασία. Ε, γιατί ξέρετε δεν έχει σημασία πόσο μακρύ είναι το σκηνή, το σημαντικό είναι να δεθεί ο κόμπος. Ε, και βεβαίως έχουμε και κάποιες γεωγραφικές διαδικασίες και τυπικές διαδικασίες όσον αφορά ε, τις ε, τράπεζες οι οποίες ε, θα συμμετάσχουν. Τέλος, όσον αφορά την ταχύτητα, όσο γρήγορα και να προχωρήσουμε θα πάρει αρκετά χρόνια και επομένως η κατασκευή αυτή καθεαυτή, ακόμα και αν όλα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά τώρα, η φυσική η κατασκευή δεν θα ξεκινήσει πριν το τέλος της δεκαετίας αυτής, γιατί ξέρετε ότι ο ίδιος ο σχεδιασμός ε, παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Είχα πολλές ε, συναντήσεις ε, τον κύριο Νίντελχεμ στο Ρόζενχάιμ, ο οποίος ήταν ο πολιτικός υπεύθυνο και ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ να εκπληρώσω το ρόλο μου ως συντονιστού λόγω της απόστασης. Όσον αφορά τώρα τον νότιο άξονα, την νότια πρόσβαση υπήρξαν σημαντικές ε, καθυστερήσεις. Πρέπει να σας πω με μεγάλη ευχαρίστηση ότι την ε, περασμένη χρονιά έγινε η επίσημη έγκριση ε, όσον αφορά την δαπάνη 1,6 δις για την κατασκευή του κομματιού από τη Φορτέτσα μέχρι το Πόντε Γκαρντένα και ελπίζουμε ότι η φάση αυτή θα ολοκληρωθεί ε, γρήγορα και επομένως ε, σύντομα θα υποβληθεί ε, η πρόταση προς αναζήτηση αναδόχων. Το σημαντικό σημείο εδώ ήταν να υπάρξει η δέσμευση κατασκευής κατά τμήματα λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες οικονομικής λιτότητας, αντί να ζητήσουμε από τις αρχές την κατασκευή ενός μεγάλου κομματιού, προσπαθήσαμε, προτιμήσαμε μάλλον να κατακαιρματίσουμε ε, την ε, διαδικασία και επομένως έτσι ήταν πιο εύκολο να γίνει ε, αποδεκτή. Επίσης, να κάνω και μία παρατήρηση άλλη όσον αφορά τον νότιο άξονα, να πω ότι Έγινε πολλή δουλειά ε, μεταξύ της Αυστρίας ε, και της ε, Ιταλίας και ο κύριος Μάουρο Φαμπρίς, ο οποίος ήταν ο συντονιστής εντός της Ιταλίας, βοήθησε τα μάλα. Και νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να έχουν έναν τοπικό συντονιστή. Τελικό μου σχόλιο κύριε Πρόεδρε είναι ότι έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση πολύ μεγάλου κομματιού υποδομής ε, και έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες ε, για την εκκίνηση του, του, ε, της σύραγγας στον Πρένερο και επομένως έχουμε και αυτή τη στιγμή και στον Πολτζάνο προχωρήσει καλά και επομένως οι συμφωνίες υπάρχουν. Τώρα το κομμάτι που συνδέει την ε, Γερμανία, την Αυστρία και την Ιταλία. Εκεί έχουν συνεργαστεί και τα επιμελητήρια και οι δήμαρχοι. Πέρα από τα τεχνικά ε, ζητήματα που αφορούν την μηχανική και τις κατασκευές. Το σημαντικό είναι η ικανότητα επικοινωνίας και νομίζω ότι το μάθημα που μαθαίνουμε από αυτή τη συνεργασία είναι ότι δεν είναι δυνατόν ε, να, ε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κινητοποιηθούν όλοι και πρέπει να κινητοποιούμε διαρκώς, να κρατάμε επαφές, να κρατάμε όλο τον κόσμο σε επαφή μεταξύ του γιατί διαφορετικά πραγματικά ξεχνιέται πάρα πολύ εύκολο. Ε, ξεκινήσαμε και ένα διάλογο με, το, με την ε, συνθήκη του ε, Alt Plain, ε, με τους δημάρχους δηλαδή της περιοχής, έτσι ώστε να δούμε μαζί τους όλα τα ζητήματα των διάβλων των Άλπαιων. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω ότι κάναμε σημαντική πρόοδο, καταφέραμε να βρούμε και λύσεις για τους παράλληλους δρόμους, Έχουμε ήδη οργανώσει την εκτέλεση της υποδομής και αρχίζουμε να δουλεύουμε για τα λεγόμενα συνοδευτικά μέτρα. Και ξέρετε ότι για να μεταφερθεί ε, ο όγκος των μεταφορών, να μετακινηθεί από το δρόμο στις σταθερές τροχιές, χρειάζονται και συνοδευτικά έργα. Βεβαίως ακόμα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τι ευχαριστίες μου στον Λέο Χούμπερς της ε, Κομισιόν που με τον επαγγελματισμό του και την αποτελεσματικότητά του ήταν πάντα πολύτιμος παραστάτης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόξ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, δύο λεπτά αυστηρότατα και αυτά είναι δύο λεπτά του, της Βορείου Ευρώπης, ο κύριος Καντσιάν για το ΕΛΚ. Ναι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πατ Κόξ, τον εισηγητή και τον συγχαίρω για αυτή την εργασία, για αυτόν τον κύριο άξονα με προτεραιότητα ακριβώ είναι σημαντική εργασία, ιδιαίτερα λεπτή και σε βραχή χρονικό διάστημα κατάφερε πολύ καλά να συντονίσει. Να τονίσω δε αυτόν τον πράσινο διάδρομο που είναι πολύ σημαντικός και θα ήθελα να ευχηθώ να πάμε πραγματικά προς την κατεύθυνση αυτή, όπως και τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία μας είπε, ώστε σιδηροδρομικά να μεταφερθεί οτιδήποτε είναι δυνατό το κύριο σημείο είναι η σύραγγα αυτή, αυτό το πολύ σημαντικό σημείο γιατί είναι στη μέση ακριβώς αυτού του διαδρόμου. Και το cross financing είναι πολύ σημαντικό γιατί συζητήσαμε ιδιαίτερα το τι μπορούσαμε να πάρουμε από την Α22, από τον Α22 Διεθνή Δρόμο που έχει προκήρυχθεί για παραχώρηση και με τη δυνατότητα στο Βερόνα Φορτέτσα να επενδύσουμε γιατί έχουμε μόνο τη σύραγγα και δεν κάνουμε και τα υπόλοιπα στη σύνδεση ε, εκεί που συνδέει αυτά τα σημεία στην Ευρώπη ε, δεν θα ε, κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, αλλά θα, μείνουν, θα την αφήσουμε στη μέση. Και επίση για τον συντονιστή, ε, για πέντε εβδομάδε ε, το επόμενο καλοκαίρι για τη συντήρηση στο Βορρά σχεδιάζουν να κλείσουν αυτό το διάδρομο. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο λεπτό σημείο, χρειάζεται να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση σχετικά με αυτό, γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχιση τη εργασία σα. Ευχαριστώ ο κύριο Καντσάν, ο οποίος ε, κάλυψε ακριβώς δύο λεφτά. Ο κύριος Σάρτελ για το ο, τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Όπως με ακούτε είμαι από τη Βαβαρία, οπότε και μένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερο το τμήμα της ε, ε, οδού αυτής ε, που είναι στη χώρα μου και βαίνει προς την Αυστρία. Ξεκινώ από το Μπρένερο. Ξέρετε ότι έχει γίνει μία μελέτη στο τετράγωνο από την εταιρεία Ράσλερ όπου λέγεται ότι δεν θα ε, μπορέσει να προχωρήσει διότι δεν θα υπάρχουν πόροι. Γνωρίζετε αυτή τη μελέτη και πώς την αξιολογείτε. Δεύτερον σχετικά με το ΕΑΤΜΕΣ e δηλαδή το κομμάτι Μόναχο Βερόνα ε, έχει προβλέψει μια χρηματοδότηση 38 δις και όπως ελέγχθη ε, πρόσφατα ε, πρόκειται να υπάρξει μία εναλλαγή η οποία να είναι λιγότερο δαπανηρή ε, δηλαδή εξαφανίστηκε η χρηματοδότηση ή πού θα πάνε τα χρήματα αυτά. Είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Έχω δύο ερωτήσεις προς το παρόν για να μπορέσω να περιοριστώ στα δύο μου λεπτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κιούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω στον κύριο Κόξ θερμά διότι ε, τα δύο τούνελ αυτά του Μπρένερο τα έχει επεξεργαστεί όπως το έπραξε διότι πρέπει να δούμε πώς θα αντεπεξέλθουμε ε, στα εμπόδια που υπάρχουν από πλευράς χώρου διότι αν κοιτάξουμε ε, το τωρινό τούνελ ε, την τωρινή σύραγγα υπάρχει ένα πραγματικό διέξοδο στο συνδυασμό οδικής διελεύσεως και τρένου και ε, ξέρουμε ότι με το Λέσμαχ ε, και το Σανγκοτάρ προς Ρότερνταμ υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία δίωδος από την Ιταλία προς τη Γερμανία και είναι καλό ότι τώρα μπορεί μπόρεσε να υπάρξει συνεννόηση με τον Γερμανό Υπουργό Δημοσίων Έργων ε, για να, και Μεταφορών για να δούμε πόσο θα μπορέσουμε να συνδεθούμε και να προωθήσουμε τις προτεραιότητες αυτές για να συνδεθούμε και με τις Σκανδιναμίες. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρκερ ε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πατ Κόξ για τον ρόλο που έχει αναλάβει που δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των συντονιστών. Γιατί βλέπετε ότι πρέπει έτσι να υπάρχει μία εγγύηση για την σωστή μακροπρόθεσμη πρόβλεψη και να μην υπάρχουν και καλυμμένα σχέδια διότι ξέρουμε ότι καταρχήν πρέπει να υπάρξουν προσφορές οι οποίες μετά θα χρησιμοποιηθούν μας βοηθούν αυτές οι, με... αυτές οι μελέτες που έχουμε δεν θα μας βοηθήσουν αυτή τη στιγμή αλλά η μελέτη για το... τη σύραγγα του Μπρένερ θα μας βοηθήσουν μόνο εάν μπορέσουν να γίνουν τα έργα υποδομής βορείως και νοτίως της σύραγγος διαφορετικά είναι χρήματα τα οποία πετάμε από το παράθυρο. Γνωρίζετε γιατί έχουμε ε, καθυστερήσει. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ξέρουμε ότι η Βόρεια υπάρχουν προβλήματα, ε, καθυστερούμε ακόμη στον προγραμματισμό και θα ήθελα να μου πείτε πόσο ε, έχετε εσείς αξιολογήσει στη συνεργασία και στις συζητήσεις που έχετε με τον Υπουργό Σάουερ πώς θα προχωρήσουμε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση Τη της συνδέσεως από γερμανικής πλευράς όντως να ολοκληρωθεί. Ο κύριος Κράμερ τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα να έρθω και ζητώ και πάλι τον λόγο αλλά ο συνάδελφός μου με ενημέρωσε. Ο, ο διάδρομος είναι Βερολίνο προς Παλέρμο και ανατολικά προς το Όσλο, Κοπενχάγη ε, και ε, ε, στο Χόλμη τι μέλη γενέστε θα υπάρξει συνέχιση αυτή προς τη Στοκχόλμη μέσω Ροστόκ και θα ήθελα να ρωτήσω υπάρχει κάποια εγγύηση από την Ιταλία ότι θα επενδυθούν αυτά τα χρήματα ε, για την νότια πλευρά του Μπρένερ ή πρόκειται απλώς για δηλώσεις και τι θα γίνει με τις εμπορευματικές μεταφορές γιατί από ό,τι ξέρω ε, η σύραγγα του Μπρένερ δεν ε, ενδείχνεται για τις εμπορευματικές μεταφορές οι οποίες θα παραμείνουν στην παλιά σύραγγα θα ήθελα σχόλια της Ιταλίας αυτά. Μετά άκουσα ότι η γέφυρα της Μεσίνας έχει ακυρωθεί. Έχετε ενημέρωση από την Ιταλική κυβέρνηση, γνωρίζετε τι έχει γίνει. Είχε ήδη ακυρωθεί μία πρώτη φορά διότι η Γερμανία είχε προτείνει μία διαφορετική λύση για όλη την Ευρώπη και θα ήθελα να ξέρω πώς πώς επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, διότι δεν μπορεί να αφήσει ένα, ένα, τη κυριαρχία ένα κράτος να υπογράφονται συμφωνίες και να μην γίνονται σεβαστές. Τι κάνετε εσείς και τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, εγώ προς τον κύριο Κόξ ακολουθώ αυτά που είπαν και οι προλαλήσαντες και όλα αυτά είναι σε συνδυασμό, δηλαδή το θέμα του προσπαθώ να σας εκφράσω διπλωματικά ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη Γερμανία για την σύναψη συμφωνιών οι οποίες δεν γίνονται σεβαστές. Δεν θέλω εδώ να δημιουργήσω ένα καυγά, αλλά, γερμανικά, ε, ε, αλλά γεωγραφικά η Γερμανία είναι κρίσιμη και ε, από ό,τι άκουσα θα συναντηθείτε με τον Υπουργό Ραμσάουερ για να υπογράψετε κάποια συμφωνία για την Αυστρία. Είναι θετικό και ένα καλό πρώτο πρώτο βήμα. Αλλά θα σας έλεγα ότι η Γερμανία στο παρελθόν έχει υπογράψει πολλές συμφωνίες τις οποίες δεν σεβάστηκε. Οπότε θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις επεμβάσεις και όσον αφορά το θέμα του πράσι, της πράσινης σύραγγας για τον Μπρένερο και τη σχετική ομάδα εργασίας. Έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες και δεν θα αναφερθώ εδώ λεπτομερώς. Πλην όμως η χρήση του τούνελ για την διέλευση άλλων ενεργειακών πυρηγών και άλλων διασυνδέσεων γεωθερμικών τα, τη διοξιδίου του άνθρακος δηλαδή έχει αξιολογηθεί ο ρόλος των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος για τον Μπολζάνο ε, ε, πολλά πράγματα που δεν αυτεπάγγελτα αλλά πρέπει να υπολογιστούν και ε, να εκτιμηθούν με πιλωτικά προγράμματα. Όπως είπατε, είναι ένα βασικό μέρος της οικονομικής συνδρομής. Ε, υπάρχει το θέμα της Ιταλίας, το οποίο ε, αναφέρατε, που προβλέπει να θέσει σε μειοδοτικό διαγωνισμό για ανάθεση σε μία εταιρεία για δεκαετίας των διοδίων πράγμα το οποίο θα επηρεάσει το πρόγραμμα και θα το επιβαρύνει με 1,5% 1,5 ε, ε, δισεκατομμύριο ε, επιπλέον χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο είναι πολύ βαρύ. Όσον αφορά το κλείσιμο της γραμμής για συντήρηση το καλοκαίρι, είναι κάτι το οποίο γνωρίζω γιατί σαν συντονιστή όπου πηγαίνω είναι το πρώτο που μου λένε είτε πρόκειται για την Αυστρία είτε για άλλες χώρες μας είπαμε πόσο αντιπαραγωγικό είναι αλλά αν δεν γίνει τότε ενδέχεται να υπάρχει με πιο μακρά περίοδος καθυστερήσεων και δεν θα ξέρουμε πότε θα σταματήσει. Δεν μπορώ να επηρεάσω την έκβαση αυτού του θέματος αλλά έχει σημασία ιδίω για τους επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σχετικά σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Χέρτοκ θα ήθελα ένα αντίγραφο διότι δεν γνωρίζω αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη που αναφέρατε ε, σχετικά με την οικονομική μελέτη και ευχαρίστως να τη δω για να την αφισβητήσω και έτσι θα μπορέσω ίσως να βρω την δυνατότητα στο άμεσο μέλλον να, να παρουσιάσω μία άλλη εναλλακτική οικονομική λύση. Ε, όσον αφορά την ε, Βερόνα ε, και τη Γερμανία, οι Ιταλοί θέλουν να αναπτύξουν ένα πράγμα και η Γερμανία άλλο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα εθνικής βιομηχανικής πολιτικής αλλά ε, επεμβαίνουν πολλές ε, δυνάμεις και το έχω συζητήσει με συντονιστές ε, στη Γερμανία φέτος το Μάρτιο στο Βερολίνο με τον κύριο Ραμσάουερ και με εντυπωσίασε ότι σε τις περισσότερες συζητήσεις μας στο διάλογο μπορούμε να συνοψίσουμε τις απαντήσεις με μία λέξη. Όχι. Λοιπόν, ε, δεν νομίζω ότι αυτό έχει σχέση μόνο με τα δίκτυα αυτά, αλλά γενικότερα, διότι εκτός από το παράδειγμα αυτό διαπιστώνουμε ότι το σύστημα αυτό, αυτό καθεαυτό τα Υπουργεία, το πολιτικό επίπεδο πάσχουν ακόμη από τις επιπτώσεις του προγράμματος του Τγκάρδη 21 και ε, ε, επηρεάζει αυτό και ε, είναι εις βάρος όλων των μακροπροθέσμων προγραμμάτων και αυτό που ελέγχθη εχθές όντως ισχύει. Πρόκειται να διατυπωθεί μία δημόσια πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα είναι καινοτόμα ε, και ποιοτικά και θα μετακινηθεί προς το καλύτερο αν μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση το Κοινοβούλιο να έχει δικαίωμα συναποφάσεως και να μπορέσει και το Συμβούλιο να ξεμπλέξει το κουβάρι. Ε, ε, ε, αλλά τότε το Κοινοβούλιο θα μπορέσει μετά να πλέξει ένα σωστό στόχο. Αυτό το αναφέρατε πολύ από εσά. Και όσον αφορά το βόρειο άξονα και τη γερμανική πλευρά, σας είπα τι προβλέπετε για το Ρόζενχάιμ για τον Ιανουάριο και ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό ε, είναι ένα κοσμοϊστορικό πρόγραμμα που θα αλλάξει τον κόσμο αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια όπου εμφανίζονται διάφοροι δημόσια για να προσυπογράψουν το συντονισμό και αυτό είναι ένα βήμα προς τα εμπρός γιατί μέχρι στιγμής ήταν όλοι διστακτικοί και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιτύχουμε όχι μόνο τα Υπουργεία αλλά και οι εταιρεία αεροδρόμων και η γερμανική DB η οποία προβαίνει στον προγραμματισμό των σιδηρονόμων έχω κάνει συζητήσεις άτυπες με το DB και ε, ε, ε, μας είπαν ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί σε χαμηλότερο κόστος από αυτό που προέβλεπε το γερμανικό πρόγραμμα υποδομών οπότε έτσι έχει και πιθανότητες περισσότερες να εγκριθεί. Αλλά όσον αφορά τα βήματα τα οποία θα αναλάβουμε <coughs> χρειάζομαι την καλή θέληση αυτής της Επιτροπής αλλά και την πολιτική καθοδήγηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά τα περιβαλλοντολογικά προγράμματα σε τόσο περιορισμένο χρόνο. Πρέπει να σας πω ότι όταν μιλάμε για την επικοινωνία, η επικοινωνία είναι διμερής και περιλαμβάνει και την ομιλία αλλά και την ακοή. Πρέπει να ακούμε καλύτερα για να προλαμβάνουμε καλύτερα τις ανησυχίες των κοινοτήτων και να τις διασκεδάζουμε. Σας είπα τι γίνεται στο Ιταλικό-Αυστριακό τμήμα του διαδρόμου ε, ε, ότι είχαμε ένα πολύ καλό διάλογο. Αν μπορώ να κάνω το ίδιο και στη βόρεια πλευρά προς τη Γερμανία δεν θέλω να υπάρξουν εκπλήσεις, θέλω να μπορέσουν οι κάτοικοι να είναι περήφανοι για αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα την Ιταλία, ναι, ε, η ερώτηση είναι ότι οι δεσμεύσεις που έχω όσον αφορά τη σύραγγα του, ε, Μπρένερ, ε, του Μπρένερο, καθώς επίσης και το κομμάτι Φοντέτσα Ποντεγκαρντένα, είναι συγκεκριμένες δεσμεύσεις και έχουν ήδη εγκριθεί από την Υπουργική Επιτροπή Δαπανών και από τον ίδιο. Ε, ε, μπορεί να γίνει μέσω αλλαγής ε, του νόμου του, της Ιταλίας, του οικονομικού νόμου της Ιταλίας έτσι ώστε να γίνει δεκτός ο κατακαιρματισμός του έργου και επομένως η κατασκευή του κατά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο ε, ε, Α22, έχουμε ήδη μία οικονομική δέσμευση της τάξης των 44 εκατομμυρίων έτος και επομένως ε, πρόκειται για μία συγκεκριμένη δέσμευση. Βεβαίως τώρα έχουμε μία νέα κυβέρνηση στη Ρώμη και βεβαίως θα ήθελα να ξεκινήσω διάλογο μαζί τους. Όσον αφορά τώρα την σταθερή ζεύξη των ε, στενών της Μεσίνης, ε, <clears throat> τη γέφυρα δηλαδή αυτή, ε, αυτό μάλλον είναι θύμα των μέτρων λιτότητας. Εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει να σας πω ότι οι συζητήσεις όπως ήταν και για τον Μπρένερο και για την Μεσίνα είναι συγκεκριμένες. Ε, για το NTMS, το συζητήσαμε αυτό. Επίσης να σας πω ότι αυτό το ε, πρόγραμμα προτεραιότητας 1 ε, θα έχει το όνομα λεωφόρος, ή διάδρομος μάλλον, υπαριθμών 5, που θα φτάνει, θα περνάει από την Ιταλία και θα φτάνει και μέχρι την Μάλτα και βεβαίως ε, αυτά πρόκειται, ε, ε, αυτό είναι σχέδια για το μέλλον, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση, ένας άξονας Ανατολής Δύσης και όντως θα πρόκειται για έναν άξονα ο οποίος θα διασχίζει από Δυσμάς προς Ανατολάς την Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Περνάμε στον επόμενο συντονιστή, εσωτερικές πλωτές οδοί ε, προγράμματα προτεραιότητας 18 και 30. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κάρλα Πέις. Uh, Κάρλα, έχεις το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν. Uh, Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Οι εσωτερικές πλωτές οδοί κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος ε, στην ε, Ευρώπη. Ξεκινήσαμε από πολύ μακριά και τώρα πλέον μιλάμε για εσωτερικές πλωτές οδούς ε, οι οποίες είναι ισότιμες πλέον με τις λοιπές οδούς. Εγώ ως συντονίστρια κυρίως εστιάστηκα σε δύο πολύ σημαντικούς διαδρόμους, τον ε, PP18 και τον PP30. Θα ξεκινήσω με τον 18. Πρόκειται για τον άξονα ανάμεσα στον Ρήνο, Μοζέλα, τον Μέιν και τον ε, Δούναβη. Και φτάνει λοιπόν από το, Άμστερνταμ, από το Ρότερνταμ μέχρι την ε, Κωνσταντσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω ότι πολλά πλοία θα ξεκινήσουν από το Ρότερνταμ με τελικό προορισμό την Κωνσταντζα, γιατί υπάρχουν και άλλε εναλλακτικέ λύσει. Αλλά ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό διάδρομο. Πρώτον, γιατί περνάει από πάρα πολλέ χώρε, οι οποίε ε, παρουσιάζουν πολιτικέ ιδιαιτερότητε, ε, διαφορέ μεταξύ του, κυβερνητικέ αλλαγέ, αλλαγέ δηλαδή στι κυβερνήσει, και ε, επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Δεν μπορώ να πάω σε μια χώρα χωρίς να συναντήσω τον Υπουργό γιατί φαντάζομαι τι θα έλεγα εγώ εάν κάποιος άλλος το έκανε αυτό στη χώρα μου. Και επομένω έχουν δίκιο ότι πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή με του υπουργού. Και αν έχουμε νέο υπουργό, ανοίγει καινούριο κεφάλαιο στι επαφέ και στι ε, επικοινωνίε. Αν υπάρχει καινούργια κυβέρνηση εξ ολοκλήρου, ακόμα περισσότερο. Ε, με το σχέδιο προτεραιότητας 18. Λοιπόν, τι συγγίνεται με το διάδρομο αυτό. Στις 24 ε, Ιουνίου το Συμβούλιο ενστανήθηκε στατιστική σχετικά με την στρατηγική του Δουνάβεως. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία, διότι ο Δούναβή αποτελεί τη σπονδυλική στήλη τη στρατηγικής αυτής και δεν δεν αναφερόμαστε μονάχα στον ίδιο τον ποταμό, αλλά σε ολόκληρη τη λεκάνη του ποταμού. Επομένως, ε, προσπαθούμε να δούμε ε, προσπαθούμε να δούμε λοιπόν όλη την, ε, και την αυσιπλοεία αλλά και τα γύρω, δηλαδή την αποφυγή πλημμυρών, την γεωργία κτλ. Πρόκειται λοιπόν για πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις τις οποίες εμείς βλέπουμε με έναν ολιστικό ολοκληρωμένο τρόπο. Υπάρχουν ε, κάποια κρίσιμα κομμάτια και ε, στρέφομαι άμεσα ε, προς τους κύριους Κράμερ και Χέρτσοκ γιατί γνωρίζουν τα προβλήματα αυτά. Ξεκινούν, ξεκινά λοιπόν μία ε, μελέτη μαζί με την ε, Επιτροπή Εποπτείας. Έχει ξεκινήσει μάλλον και προοδεύει. Η πρώτη ενδιάμεση αξιολόγηση, μάλλον η πρώτη ενδιάμεση αναφορά θα γίνει το Δεκέμβριο. Η Επιτροπή ε, στο εσωτερικό της δουλεύει με πάρα πολύ καλό και αρμονικό τρόπο και σε γενικές γραμμές υπάρχει συμφωνία. Η Επιτροπή Εποπτείας, λοιπόν, Monitoring Committee, ε, ε, είναι μια επιτυχής ε, διαδικασία και όλες οι ενδιαφερόμενες και εμπλεκόμενες χώρες έχουν εκπροσώπους. Το 2012 αναφέρουμε, περιμένουμε μάλλον να μένουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση ε, για την εσωτερική κυκλοφορία. Άκουσα προηγουμένω τον κύριο Χέρτσογκ να λέει ε, ότι η διασύνδεση Γερμανίας-Αυστρίας είναι ε, μία περιοχή με υπερβολικά μεγάλη κυκλοφορία και αυτό λοιπόν νομίζω ότι η διάνοιξη θαλασσία, συγγνώμη, πλωτών εσωτερικών οδών μπορεί να αποσυμφορήσει την υπερβολικά συμφορημένη αυτή περιοχή. Uh, και επομένως ε, ε, κάνουμε και προσπάθειες ε, να προβλέψουμε ποια θα είναι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από από την μετακίνηση ε, της ε, κυκλοφορίας προς τις ε, πλωτές οδούς. Αυτό, τα αποτελέσματα της εκθέσεως θα είναι στη διάθεσή μας το 2013 του 2012, αλλά ήδη όπως σας είπα το Δεκέμβριο θα έχουμε μία πρώτη εκτίμηση είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε τις απόψεις που έχουν οι διάφορες εμπλεκόμενες περιφέρειες γιατί υπάρχουν και κάποιες διστάμενες απόψεις και είναι σημαντικό να ε, ακουστούν όλες οι πλευρές. Τώρα, ανατολικά της Βιέννης εκεί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του Δούναβη. Βεβαίως, ερχόμενοι από την ε, Γερμανία, φτάνουμε σε, ένα πάρα πολύ κρίσιμο, ε, σε μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή ε, του ποταμού γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τη διασύνδεση Ρήνου, Μέιν, ε, Δούναβη ε, και είναι το κομμάτι που προχωράει προς την Βιέννη. Ε, η Ανατολική Βιέννη με το Εθνικό Πάρκο, σημαντικό κομμάτι, αλλά έχει καθυστερήσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επομένως έχει αυτή τη στιγμή σταματήσει, αργοπορεί το έργο. Μετά φτάνουμε στο τμήμα της Ουγγαρίας, ε, προωθείται, προχωράει η μελέτη εκεί, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση παραμένει πολύ ευάλωτη. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η Ουγγρική κυβέρνηση όσον αφορά την επικοινωνία με τον κόσμο. Αλλά ε, εξακολουθούν να υπάρχουν ε, κάποιες καθυστερήσεις και το θέμα είναι να προχωρήσει η μελέτη χωρίς ε, καμία ε, παρίσφρηση της ε, κυβέρνησης. Βουλγαρία, Ρουμανία και εκεί εκκρεμούν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο συνολικός συντονισμός δεν είναι εξαιρετικός, δεν είναι τέλειος, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι μπορούμε να βελτιωθούμε εδώ. Στο Καλαράζι υπάρχει μία ε, αργοπορία όσον αφορά το πρόγραμμα εποπτείας. Τώρα αυτό το πρόγραμμα, το monitoring program έχει συμφωνηθεί. Και ε, επίσης οι ορνηθολογικές μελέτες ε, ολοκληρώνονται. Έχουμε δείγματα ε, ε, έχουμε δείγματα ζωής συγκεκριμένα. Επίσης έχουν μπει ε, πομπή σε 30 είδη έτσι ώστε να παρακολουθηθούν οι διαδικασίες. και επίσης έχουν μπει πομπή και σε ψάρια τα οποία ε, θα ε, παρακολουθηθούν. Δεν φαίνεται να του ενοχλεί καθόλου ο πομπό αυτό. Εν πάση περιπτώσει ε, έχουν, θα αρχίσουν γρήγορα οι εργασίες γιατί θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν και περισσότερο Υπάρχουν και περισσότερα προγράμματα, μικρότερα, αλλά το ε, πρόγραμμα 30 είναι πολύ σημαντικό, διότι για πρώτη φορά θα είναι δυνατόν να ε, μπορέσει κανείς να συνδέσει τη, από την Βόρειο Θάλασσα μέσω των καναλιών τη Γαλλία ε, στο Ρότερνταμ και στην Νόιζε. 5 Απριλίου 2011 ήταν ένα πολύ βασικό γεγονός διότι ξεκίνησε μέσω του Προέδρου Σαρκοζή ε, ο διάλογος για τη δημιουργία του καναλιού αυτού το οποίο ε, θα ολοκληρωθεί εντός 15 μηνών και περιμένουμε ότι στη συνέχεια ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά αυτή ήταν η δέσμευση της γαλλικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, όλα αυτά είναι κάτι το οποίο προχωρά και ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε βάσει του σημαντικού προγράμματος το οποίο έχει ξεκινήσει και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει ε, μία διακυβερνητική επιτροπή και καταφέραμε να εμπλέξουμε και την κυβέρνηση της Ολλανδίας και της Γερμανίας εάν το επιθυμούν. Ε, δηλαδή ε, ε, εφ' προσκαλούνται σε όλες τις συνεδριάσεις και αυτό είναι σημαντικό διότι πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το κόστος των διοδίων για όλη την διέλευση ε, και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες για την επιτυχία του διάβλου. Ε, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το πρόγραμμα και ε, θα πρέπει να δοθεί μία μορφή η οποία ε, να συμβάλλει στην επιτυχία αυτής της διάβλου. Γι' αυτό και ε, κάλεσα ε, τον κύριο Κάλλας και τον κύριο Σαβαρή στην Βουδαπέστη όπου συζητήσαμε με τις διάφορες ε, με τα διάφορα μέσα που θα συμμετείχαν και ε, από για τη Μάντοβα υπάρχει ε, από τη Βενετία μέχρι τη Μάντοβα ε, ο κύριος Καστέλη, ο κύριος Καντσιάν και άλλοι συνάδελφοι όπου συζητήσαμε για μια νέα λύση η οποία θα παρακάμψει το βεβαρημένο σύστημα της περιοχής και ελπίζω ότι έχουμε καλές πιθανότητες να μπορέσει να υπάρξει μία επέκταση μέχρι το Μιλάνο, πράγμα το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για αυτή την περιοχή, για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στους αυτοκινητοδρόμους, ε, όχι ίσως για τα φορτηγά, αλλά για τα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ Κάρλα, με συγχωρείς ε, που πιέζουμε αλλά προσπαθούμε να προωθήσουμε το θέμα. Βλέπω ότι τώρα έχουμε 7, 2 ε, λεπτά και θα πατάω το κουμπί μόλις υπερβαίνετε τα 2 λεπτά για να έχετε μια ευγενή παρακολούθηση. Ο κύριος Μαρινέσκου. Ναι, αγαπητέ συνάδελφοι, εσείς παρουσιάσατε αυτό το σχέδιο του Δούναβη, μιλήσατε για το Ρήνο, μιλήσατε για τη στρατηγική νομίζω για τον Δούναβη που είναι πολύ σημαντικό κείμενο και πέρα από την αυσιπλοεία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Αλλά στο τέλος ε, της όλης ιστορίας. Εάν αυτός ο διάδρομος δεν είναι για τις μεταφορές, τότε οι υπόλοιπες πτυχές δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο διάδρομος αυτός που θα συνδέει την Κωνσταντσα με το Ρότερνταμ να αποτελέσει ένα διάδρομο σημαντικών μεταφορών για την Ευρώπη. Να έχει δηλαδή ευρωπαϊκή σημασία. Τώρα αναρωτιόμαστε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτός ο συντονισμός για τη στρατηγική του Δούναβη. Εκεί προβλέπονται αρκετές πτυχές και σε κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά συμμετέχουν και συντονίζουν δύο κράτη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς θα γίνει ο συνδυασμός ε, και συνεργασία αυτών των συντονιστών. Ε, αυτά τα προγράμματα τα οποία προωθούνται και που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτόν το διάδρομο σε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα γίνει η σχετική διαχείριση. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ναι, τα πράγματα πραγματικά προχωρούν. Αυτό καταλάβαμε από όσα μας είπατε. Το 18 ε, θα μιλήσει ο συνάδελφος από την ομάδα μου. Είναι περίπλοκο. Ακούσαμε μια λεπτόμερη περιγραφή τώρα για το σχέδιο αυτό έχει τρομερές δυνατότητες. Έχει να κάνει με το Βέλγιο, των Ολλανδία, την περιοχή του Παρισιού και με τη Γερμανία και ε, τη συνδυασμό με το σχέδιο 18. Μας υπενθυμίσατε στη συνέχεια ότι η σημασία αυτής της διαδρομής ποια είναι και επίση τα διόδια. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά αλλά και ευαίσθητα. Γνωρίζουμε ότι τα έργα αυτά κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα, χρειάζονται την κατάλληλη χρηματοδότηση και μέσω των διοδίων. Αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε πώς, ε, πώς θα καθοριστούν αυτά τα διόδια, ποιο θα είναι το ύψος τους, να αποφύγουμε προστατευτικές πολιτικές, να αποφύγουμε ένα ανταγωνισμό που με δυσκολίες ίσως υπάρξει μια αποθάρρυνση για την χρήση αυτών των νέων δρόμων και ίσως συνεχίσουν ε, μέσω ε, μεσοϊδάντινης διαδρομής. Ποιος θα αποφασίσει η Γαλλία, ας πούμε, τι γίνεται, ποιος θα συντονιστεί, πώς θα συμμετέχει. Θα ήθελα να γνωρίζω μερικά πράγματα περισσότερο όσον αφορά τα διόδια. Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λοιπόν, ε, πρόκειται για ένα από τους τομείς τους πιο πράσινους ε, με τις ε, ενδοποτάμιες ακριβώς οδούς και σχετικά με το σχέδιο 8 και τον έλεγχο τη σχετική επιτροπή, η οποία ασχολείται με κάθε πτυχή, ακόμα και με τη δυνατότητα του να μην γίνει τίποτα, μέχρι την πιο ευρία δυνατότητα, δηλαδή να έχουμε πάρα πολλά έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν. Τι γίνεται ακριβώς, συγκεντρώνεται κανείς σε ορισμένα μέρη που θα μπορούσαν να συνδυαστούν, τι γίνεται και ακόμα η Επιτροπή Ελέγχου έχει διδαχθεί κάτι από τη σύνδεση ε, του Δούναβη έχει ωφεληθεί. Και στην έκθεση την Μπέγκιν ε, νομίζω ότι μιλήσαμε αρκετά για τη φύση. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς, αν θέλει κανείς ε, να πάει με ποδήλατο, ε, διαπιστώνει ότι δυστυχώς σε μια περιοχή φυσικού κάλους έγινε μια επέμβαση. Όλα αυτά η Επιτροπή τα εξέτασε, διδάχτηκε από την, ε, από την περίπτωση αυτή του Δούναβη. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ, <clears throat> ευχαριστώ. Θα περιοριστώ λόγω του χρόνου σε ένα σημείο που αναφέρεται στο τμήμα ανατολικά της Βιέννης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε προσπαθήσει να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις και ε, να μην ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις για την κατάρτιση ενός εθνικού πάρκου και γι' αυτό τα πράγματα στράβωσαν. Είναι κάτι λοιπόν που δεν θα διορθωθεί τόσο γρήγορα. Λοιπόν πρέπει να δούμε μήπως μπορεί κάτι κάτι να γίνει με τα οχήματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά διότι δεν είναι υποχρεωτικό να αναλυφθούν μόνο οικοδομικά μέτρα αλλά υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία θεωρώ πιο αποτελεσματικά για την προώθηση της οδικής επικοινωνίας π.χ. η γραφειοκρατία με την Σερβία η οποία δημιουργεί τρομερά προβλήματα. Γι' αυτό και εδώ θα έπρεπε να δούμε ακριβώς τι προσφέρεται και δεύτερον σχετικά με τα πλοία τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο Δούναβι πρέπει να είναι γιγαντιές οι επενδύσεις για να μπορέσουν να διορθώσουν τα στραβά. Γι' αυτό και δεν προχωράμε τόσο γρήγορα Ίσως ε, θα έπρεπε να γίνει κάποιο πρόγραμμα με προσαρμοσμένα σκάφη γιατί τώρα αν ονειρευόμαστε απλώς και περιμένουμε υπομονετικά δεν θα πετύχουμε κάτι. Επίσης πρέπει να δούμε τι είναι ε, σοβαρά τα αγαθά τα οποία μεταφέρονται εις ε, ποτάμια. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Δούναβη και παρακαλώ να το κοιτάξετε πιο προσεκτικά. Λοιπόν, ε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα την κυρία Πέις. Εδώ μιλάμε για την Άγια Μπράιλα και έχουν ε, οριστεί εργασία για τέσσερα ολόκληρα χρόνια για την ε, προστασία όλων αυτών ε, των ειδών καθώς και για άλλους ε, λόγους περιβάλλοντος. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την πραγματοποίηση αυτού το καλοκαίρι υπήρξαν πολλά προβλήματα στο Δούναβι ακριβώ επειδή υπήρξε μια κάποια αποξήρωση λόγω λιγοστών υδάτων. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, πώς μπορεί κανείς ε, να μπει στα πλαίσια αυτού του Connecting Europe. Ε, οι ε, λιμένες του Δούναβη θα έχουν ε, σημασία νομίζω και θα πρέπει να δούμε το συνδυασμό λιμένων στο Δούναβι που με τη Μολδαβία και την Ουκρανία να εγγύθουν την σύνδεση. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί ένα σημαντικό σημείο και πρόκληση για αυτό το δίκτυο και ελπίζω ότι θα υπάρξουν όσο γίνεται περισσότερα λιμάνια στο Δούναβι. Ακόμα κάτι, διάφορα κανάλια που θα μπορούσε να υπάρξει ε, που θα μπορούσαν να πλεύσουν πλοία στο Ρήνο και επίσης η προσαρμογή των στόλων των πλοιαρίων των πλοίων. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα συνεχιστούν και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ε, βοήθειά σας. Κράμερ. Ευχαριστώ. <clears throat> Ξέρετε ότι ε, για τον Ρήνο χρηματοδοτούμε ε, τα όνειρα και πιστεύουμε ότι και για το, το Δούναβι, εάν τον δημιουργήσουμε θα μπορούμε να κάνουμε κάτι. είχα πάει παλιά προετών μία κρουαζιέρα στον Δούναβη και είχα συναντήσει πολλά μεγάλα πλοία. Τώρα είδα μόνο τρία πλοία την τελευταία φορά που πέρασα, διότι υπάρχουν τρία επίπεδα. Θέλουμε να ενισχύσουμε ε, τον ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την, στις πλώες ε, των αγαθών στο Δούναβι θέλουμε ε, να κάνουμε ένα χώρο απορριμμάτων ή θέλουμε να κυκλοφορούν μεγάλα πλοία και να ασχολείται και να επενδύσουμε τουριστικά. Πρέπει να ε, αποφασίσουμε πώς θέλουμε να επενδύσουμε διότι σε τους σιδηροδρόμους προσπαθούμε ε, να ε, κινητοποιήσουμε τις επενδύσεις και να έχουμε πολύ υψηλό κόστος ενώ βλέπετε στα ποτάμια δεν έχουμε τόσες πολλές πληρωμές και ε, εάν παντού στις εσωτερικές πλώες στην Ευρώπη να υπάρχει πληρωμή διοδίων αυτό δεν θα υπάρξει χρειαζόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός και στις εσωτερικές πλώες Οπότε πρέπει να υπάρχουν και επίπεδα για τις εκπομπές και μια καλύτερη οικονομική διαχείριση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέρτουγκ, βεβαίω αντιλαμβάνεστε ότι στέλνω, απευθύνω τι ερωτήσει μου σε συγκεκριμένα θέματα. Ε, έχουμε μιλήσει για ε, το κόμμα του Μπετόν στη Βαβαρία και με ασλέγουν λέγουν ότι πρέπει να βελτιώσουμε την περιοχή. Ε, όντως έχει έτσι κατάσταση γιατί θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στην περιοχή μου και ποιος αποφασίζει η δική μας ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Πέις έχει 10 λεπτά για να απαντήσει τώρα. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μαρινέσκου. Με ρωτάτε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτόν τον ε, σημαντικό διάδρομο με τα ΔΕΔ. Κύριε Μαρινέσκου, έχει μια εντελώς νέα προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προς αυτό. Ε, δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά όσον ούπο και νομίζω ότι θα φτάσει και στο Κοινοβούλιο. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και έχετε σαφή άποψη για το τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον και ποια θα πρέπει να είναι η μελλοντική προσέγγιση των ΔΕΔ. Θα απαντηθεί αργότερα λοιπόν το ερώτημά σας. Ο κύριος Καντράουι, καντράουι. πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα διόδια. Αυτό είναι το χάμφραχ, όπως λέμε στα Ολλανδικά. Αυτό είναι ακριβώς το ψητό. Δεν είναι μόνο θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γαλλικής Κυβέρνησης, της Βέλγικης Κυβέρνησης, των δύο τμήματων ε, αλλά και η Επιτροπή των Χριστών συζητάει. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η Επιτροπή των Χριστών, γιατί αυτοί ε, μπορούν να έχουν άποψη λέγοντας ότι εάν τα διόδια εφαρμοστούν έτσι δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ, ε, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ αυτά τα κομμάτια της εσωτερικής πρώτης εάν το βάλετε το διόδιο αλλιώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Γίνεται επίσης συζήτηση στην Διακυβερνητική ε, Επιτροπή με τρόπο ώστε τα διόδια να εφαρμοστούν ε, ε, έτσι ώστε το κανάλι τελικά να χρησιμοποιείται και από τους απλούς χρήστες και από τις εταιρείε. Ε, είναι πάρα πολλά ε, τα φορτία τα οποία πηγαίνουν προς την κατάθεση αυτή ε, και πρέπει να πω ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη εξυπνάδα αυτό το κομμάτι του διαδρόμου με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο επαναλαμβάνω και πιστεύω ότι το κανάλι αυτό μπορεί να έχει εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Και στη δικιά μου περιφέρεια στις κάτω χώρες βλέπω ότι ε, υπάρχει μεγάλη κίνηση φορτίων προς την, ε, και από την Γαλλία. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι ε, μεγάλη επιτυχία. Και εάν εφαρμοστούν διόδια θα το αποφασίσουν τελικά οι ίδιοι οι χρήστες. Το χρονοδιάγραμμα σύντομα, αλλά δεν μπορώ να σας πω ε, ε, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να σκαφτεί και ολόκληρο το κανάλι, άρα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μας. Αυτά για τα διόδια. Κύριε Φαντάλε, η Monitor Committee, η Επιτροπή αυτή η Εποπτείας, κάνει τη δουλειά της. Ε, δεν μελετάει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά οτιδήποτε προκύψει από τη μελέτη σε της ε, κατασκευής των 17 χιλιόμετρων. Οποτεδήποτε προκύψει κάτι το ε, συζητάει. Ε, σας είπα και προηγουμένως ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες ήταν λίγο πεπαλαιωμένε, επομένως έπρεπε να ξαναρχίσουν. Και επομένως η Επιτροπή αυτή κοιτάει όλα τα θέματα. Το ξέραμε αυτό από πριν. Ε, και είχαμε και μέχρι το 12 για να ολοκληρωθούν ε, οι μελέτες αυτές. Το 12, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα έχουμε το αποτέλεσμα της ε, μελέτης. Και στην Επιτροπή αυτή υπάρχουν και, και από την πλευρά του περιβάλλοντος τέσσερα άτομα και από την πλευρά των, της βιομηχανίας άλλα τέσσερα ε, έτσι ώστε να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα και να μην έχουμε μετά ε, περαιτέρω διενέξεις εκ των υστέρων. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, το κομμάτι ανατολικά της Βιέννης ε, δεν κατάλαβα πολύ καλά τι εννοούσατε. Όταν αναφερθήκατε στις τροχίες των αυτοκινητών που θα πρέπει να προσαρμοστούν στο κανάλι, στο ποτάμι, παρατήρηση της Λίχτενμπέργκερ εκτός μικροφώνου. Για τα πλοία, ναι. Κυρία Λίχτεμπέργκερ, και πέρσι και πρόπερσι και ε, αντιπρόπερσι είχατε ρωτήσει ακριβώς το ίδιο, είχατε υποβάλει ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Ξέρετε, υπάρχει και η αγορά που παίζει ρόλο σε όλα αυτά. Εμείς ε, μπορούμε να, ζητήσουμε να ζητήσουμε από τους μελετητές, από τους ερευνητές να μελετήσουν το θέμα. Εμείς μιλάμε τώρα για, την, ε, για τον διάδρομο, δεν μιλάμε για το μήκος ε, του πλοίου. Εμείς θέλουμε ε, πλοία που να πηγαίνουν από την Αύρα μέχρι το τέλος του Δούναβη Κοιτάξτε, εάν τα πλοία δεν χωράνε σε αυτό το διάδρομο, δεν έχει έννοια να το χτίσουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ε, ε, ε υπάρχει μεγάλη, ανοίγεται μεγάλη ευκαιρία για τα πλοία αυτά. Από όσο ξέρω, η Ουγγαρία έχει και δικά της πλέον ε, ναυπηγή και δικά της πλοία και πηγαίνει προς τα εκεί και εν πάση περιπτώσει η αγορά θα προσαρμοστεί στον ε, διάδρομο αυτό. Ε, τι κάνει. Τι, τι Α, η κυρία Τικάου, συγγνώμη, ναι, ναι, λέει ο η κυρία Τικάου. Η Βράιλα Καλαράς, νομίζω ότι πάμε καλά εκεί. Με απασχολεί περισσότερο το κοινό τμήμα του ε, ποταμού παρά αυτό του Καλαράση. Και η δουλειά προχωράει καλά και το monitoring project ε, προχωράει καλά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το διάδρομο αυτό με τον τρόπο με τον οποίο αρχικώς ε, θελήσαμε τότε, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και αυτός ο πολυτροπικός κόμβος. έτσι ώστε να υπάρχουν αυτές οι συνδυασμένες μεταφορές και ανάμεσα και, στους, και στις τρεις μορφές μεταφορών. Ε, και είναι γεγονός ότι σε διάφορα σημεία θα πρέπει να γίνουν τέτοιοι πολυτροπικοί κόμβοι, multi-modal hubs. Και βεβαίως ε, είναι σημαντικό και στην περιοχή που αναφέρατε να υπάρχει ένας τέτοιος κόμβος. Κύριο Κράμερ, Ένας από τους στόχους μας βεβαίως είναι και ο τουρισμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός ε, και ενδιαφέρον για την ε, περιοχή και θα πρέπει οι διάφορες περιφέρειες να μπορέσουν να προετοιμαστούν ε, για να αντιμετωπίσουν και την διάσταση αυτή. Ο τουρισμός είναι μια πραγματική ευκαιρία για όλες τις παρόχθιες χώρες. Η μόλυνση είναι όντως πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την πλευσιμότητα του ρήνου Ε, γιατί ξέρετε εγώ ήμουν μια φορά στην Ήψη και είδα μόνο τρία πλοία να περνάνε. Και σαν Ολλανδέζα εμένα αυτό με σοκάρισε. Μα ναι, μόνο τρία πλοία γιατί δεν είναι, ευκ... δεν είναι πλωτός ο Ρήνος ε, ε, ο Δούναβης παντού. Επίσης με εκπλήσει πάντα το γεγονός ότι οι Ολλανδοί στην ε, χώρα μου είναι πάντα πολύ υπέρ των εσωτερικών πλωτών ε, οδών γιατί λένε ότι είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον αυτή η μορφή ε, μεταφορών. Ενώ κάθε φορά που σας βλέπω εσείς μου φέρεστε σαν να είμαι εγώ άνθρωπος που θέλει να μολύνει προσωπικά ολόκληρο το Δούναβι ενώ εγώ θέλω να είμαι ε, μέρος της λύσης ε, για την ε, απομάκρυνση της μόλυνσης από το ρήνο. Ούτε μία τρίχα της κεφαλής μου δεν θέλει να μολύνει το ρήνο. You have a truck and you go from, from Rotterdam to, uh, to Genoa, then we made road είναι σημαντικό ότι εμείς κάνουμε πάρα πολλά, παίρνουμε πάρα πολλά μέτρα, βάζουμε σηματοφωτεινούς σηματοδότες, κάνουμε ένα σωρό πράγματα έτσι ώστε οι διάδρομοι αυτοί, οι τροχιές αυτές ε, να διευκολύνονται όλο και περισσότερο. Ε, αλλά για, στο Δούναβι δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα. Ε, και νομίζω ότι όταν θα έχουν τα διόδια τότε θα γίνει κάτι και στον ε, Δούναβι και το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο ισχύει μάλλον και στα κανάλια στο Βορρά γιατί μέχρι τώρα τα περνάνε μονάχα πάρα πολύ μικρά πλοία. Αυτά τα μικρά πλοία δεν θα πληρώνουν βέβαια διόδια αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρετε ότι με τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός δεν θα φυγεί. Και τελευταία ερώτηση του κυρίου Χέρτσουκ. Μα γι' αυτό ακριβώς κάνουμε τη μελέτη, κύριε Χέρτσουκ. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση τώρα του χρόνου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Γι' αυτό ακριβώς εκπονείται η μελέτη, ε, για να δούμε τι βήματα πρέπει να αναλυφθούν έτσι ώστε να γίνει απολύτως πλωτός ο διάδρομος αυτός. Ιδού το μέγα ερώτημα. you, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πέις. Αυτό τώρα με φέρνει στο επόμενο θέμα, αλλά ήδη έχουμε καθυστερήσει 15 λεπτά. το πρόγραμμα 21 για τις, ε, ε, ε, τους αυτοκινητοδρόμους της Ασής ο κύριος Ολιβέρα. Θέλω να αναφερθώ στις ποιοτικέ αλλαγές οι οποίες έγιναν φέτος και επίσης μετά στις ποσοτικές αλλαγές μετά από την υλοποίηση των προγραμμάτων. Με συγχωρείτε κύριο Λιβέρα, αλλά σας παρακαλώ κύριοι, ε, πού είναι οι καλοί σας τρόποι. Λοιπόν, ε, υπάρχουν ουσιαστικά θέματα για, τους, ε, για τα θαλάσσια λιμάνια και τα ποτάμια λιμάνια και πρέπει να δούμε πόσο θα μπορέσουμε να μειώσουμε ε, τις, ε, τις εκπομπές, πώς θα ολοκληρώσουμε τις μεταφορές και θα εξετάσουμε ιδιαίτερα θέματα όπως είναι η ασφάλεια και η πλοήγηση στον πάγος για τη Βαλτική ε, κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να προωθήσουμε και το εσωτερικό και το εξωτερικό εμπόριο μέσω των προγραμμάτων TNT ε, ε, και γι' αυτό εμείς ε, έχουμε προσπαθήσει να λάβουμε υπόψη όλα τα θαλάσσι, όλες τις θαλάσσιες παραμέτρους αλλά και την ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων και ε, τις ποτάμιες μεταφορές οι οποίες μπορούν να ε, εξεύρουν στήριξη ευρωπαϊκή για να αναπτυχθούν. Σε σχέση με πέρσι έχουμε μία ποιοτική πρόοδο, δηλαδή βλέπουμε τώρα την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Έχουμε 12 προγράμματα τα οποία ε, καλύπτουν περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ ε, ως κατώτατο όριο και 850 εκατομμύρια ευρώ ως ανώτατο όριο. Ε, τώρα ε, το ένα πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα και προβλέπουμε ότι το κόστος θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο θα χρειαστούν δηλαδή να υπερβούν κατά 50 ε, εκατομμύρια ευρώ τον στόχο. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε και άλλα προγράμματα πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για όλη την περίοδο χρηματοδοτήσεως 2007 2013 θα ε, μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν 30 προγράμματα περίπου κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ ε, και θα μπορέσουν μάλιστα να φτάσουν και μέχρι 2 δις. Ε, αν λοιπόν υπάρχει χρηματοδότηση θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλες οι επενδύσεις, Μάρκο Πόλο, Ιντερεκ και τα λοιπά και το κόστος θα είναι κάπως υψηλότερο πράγμα το οποίο ε, σημαίνει ότι θα ξεκινήσουμε ε, τους υπολογισμούς από το 2007 για να δούμε πώς προχώρησαν. Ε, χρειάζεται όμως το 2020 να γίνει ένας απολογισμός, να δούμε πού θα βρισκόμαστε και τι έχει επιτευχθεί σε, στις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και γενικώ ε, στις μεταφορές όπως και στα ε, ολοκληρωμένα δίκτυα TNT τα διευρωπαϊκά δίκτυα διότι υπάρχουν διάφορα στοιχεία εκ των οποίων τα περισσότερα είναι διαβλή οι οποίοι πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν σύγχρονος να μειωθούν οι εκπομπές, να αυξηθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε όλα τα ευρωπαϊκά ύδατα, να αντιμετωπίσουμε ιδιομορφίες όπως ο πάγος το χειμώνα στη Βαλτική και ε, ε, να μπορέσουμε να επιλύσουμε ορισμένα από αυτά τα προβλήματα τα οποία ε, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2013 και θα πρέπει να παραταθούν ως το 2020. Ε, έχουμε ένα νέο πρόγραμμα ε, φέτος, ε, μάλλον πέραν του ενός, εκ των οποίων τρία αναφέρονται στην διαχειριστική διοικητική μέρημνα και ένα αναφέρεται στην ενδοχώρα πίσω από τα λιμάνια και το, τη σύνδεση των λιμανιών με την ενδοχώρα για, ε, έχουμε ε, λάβει ως παρατηρητήριο τη Ριγέκα χρησιμοποιώντας ε, διάφορες τεχνικές ε, πληροφόρησης και ε, αποβλέπουμε στο να δημιουργήσουμε έναν τέτοιο, μια τέτοια διάβλο μεταξύ Ροστότ και Γκένζε και έχουμε και το πρόγραμμα Μοναλίζα και το πρόγραμμα LNG που είναι πολύ ενδιαφέρον για μας έχετε το κείμενο μου οπότε θα προσπαθήσω απλώς να αναφέρω τους τίτλους για να ακολουθήσουμε ε, για να μην επαναλάβουμε θέματα τα οποία ήδη έχουν συζητηθεί ε, πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, υποδομές ιδίως στην ενδοχώρα ε, πράγμα το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη αλλά πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον να υπάρχει ε, η ανάπτυξη εξύπνων ε, υπηρεσιών υποδομών, να καταλάβουμε καλύτερα πώς θα βοηθήσουμε τον τομέα αυτό και με ενδιαφέρουν οι πιλωτικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία έμπνευση ε, θα πρέπει να προωθηθούν οι δραστηριότητες και έχουμε πολλά παραδείγματα όπου βλέπουμε ότι η πληροφόρηση έχει βοηθήσει την διεκπαιρέωση στα λιμάνια και εγώ αποδίδω μεγάλη σημασία στη βελτιωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ε, για ε, την ε, βελτίωση του ανθρωπίνου στοιχείου στην περιοχή. Αναφέρομαι είτε εις τα πληρώματα ή στους ειδικού της διοικητικής μέρημνας θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα one-stop shop για να μπορέσει να βελτιωθεί η θαλάσσια μεταφορά και ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε το Arch» για να μπορέσει να αναπτύξει τους εξοπλισμούς διότι θυμάστε ε, ε, η, μόνη, η μόνη βελτίωση που έχουμε σημειώσει είναι στα κροαζιερόπλια, σε κανένα άλλο είδος πλοίου Γι' αυτό και εγώ πρότεινα να υπάρχει μία, ένα συντονισμός στη χρηματοδότηση και επανέρχομαι ότι και εκεί θα χρειαστεί ένα one-stop shop ε, και θα ήθελα να να δω αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες είναι υπό έγκριση ε, και οι οποίες θα διευκολύνουν το έργο και τη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών γιατί ξέρετε ότι πολλές χώρες των ανατολικών συνόρων εξαρτώνται από τα δυτικά λιμάνια και θέλουν να παραλαμβάνουν ή στην ανατολική πλευρά, στη Ρωσία, στο Καζακιστάν, στην Ουκρανία, στην Λευκορωσία που μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ευρωπαϊκών λιμανιών. Υπάρχουν όπως σας είπα τέτοιες μελέτες ε, και όσον αφορά το LNG ε, με όλες τις χώρες γύρω από την ε, Βαλτική οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν ένα σύστημα για τον ε, εφοδιασμό σε όλη την περιοχή της ε, Βαλτικής με φυσικό αέριο και βλέπουν ποια θα είναι τα προσόντα από αυτή την κίνηση. Χρειάζονται όμως όπως είπα γεωστρατηγικές μελέτες για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, δεν θα μακρηγορήσω. Τα PPPs θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, σε συνδυασμό με τις ε, πόλεις και με τα φιλόδοξα προγράμματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μία ειδική σύνδεση στο τομέα των ε, τελωνίων. Τα, η τελωνία είναι περίπλοκος τομέας και υπάρχει μεγάλη πίεση. Ε, θέλουν να φροντίσουν πολλά θέματα αλλά και εμείς εξαρτόμαστε από το μοναδικό σταθμό. Δηλαδή καλό είναι να υπάρχει συνεργασία και των τελωνίων στο πρόγραμμα αυτό. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι δίνω μεγάλη σημασία στις στατιστικές και είναι καλό να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Έχουμε 7 ομιλητές ε, από εμπειρογνώμονες και ξεκινώ με τον κύριο Κανσιάν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ το συντελνιστή Ντεολιβέρο ιδιαίτερα λεπτομερής η έκθεσή του. Να ασχοληθώ με το σημείο 7 της έκθεσής του. Θα ήθελα να τονίσω τα, την όλη διάρθρωση του θέματος ε, και πώς θα συνδεθεί με τις γήινες εγκαταστάσεις ε, και το τι θα πρέπει να γίνει. Εδώ λοιπόν το πώς θα συνδυαστούν τεχνολογικά όλα αυτά ανάμεσα οι τα διάφορα στοιχεία, τα θαλάσσια, θαλάσσια ακριβώ και θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά θα βοηθήσουν αυτό το συνδυασμό και ακόμη κάτι για τους ανθρώπινους πόρους ε, και για τον στόλο. Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και συνδυάζονται με τα ναυπηγεία που αντιμετωπίζουν κρίση. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε αυτό, θα πρέπει να έχουμε και ένα προϋπολογισμό κατάλληλο και επίσης στο PPP αναφέρθηκε και εδώ νομίζω ότι μπαίνει και η χρηματοδότηση μέσω του Project Band. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο που νομίζω ότι απέδωσε καρπούς λιγότερους από αυτούς που περιμέναμε και τι περιμένετε από τα εκομπόνους που είχαμε μιλήσει εδώ ακριβώς μέσα πριν από ένα χρόνο. Σας ευχαριστώ. Κύριο αλκαντράου δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας αυτή. Ναι, καταλαβαίνω ότι εσείς επιμένετε στις ε, επενδύσεις και στις μελέτες για την οργάνωση όσο γίνεται καλύτερα του τομέα. Πάνω σε αυτό το σημείο συμφωνώ μαζί σας, είναι κάτι το ουσιώδες. Και ακόμα κάτι. Πρώτα απ' όλα, ε, ξέρετε κάτι σχετικά με τα ισχύοντα προγράμματα, τι έγινε, ε, ποια απόδοση των επενδύσεων που έχουν γίνει εκεί έχουν, ε, έχουμε διαπιστώσει και τι έγινε νομίζω ότι θα ήθελα να μας πείτε ένα μέρος της ροής εμπορευμάτων πήγε στις θαλάσσιες μεταφορές και ακόμα σε περιφερειακό επίπεδο για τα σχέδια που έχουν επιλογή τι ακριβώς συμβαίνει και η Βόρεια Ευρώπη εκεί αποδίδεται σημασία. Πεστε μας, έχει σημειωθεί μια κάποια εξέλιξη. Υπάρχουν και φορείς στο Νότο που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες αυτές προσφέρονται. Και ακόμη, για τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθορίσει για τη μελλοντική περίοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν και το σχέδιο αυτό πώς το εκτιμάτε, λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις που γίνονται σε αιτήσια βάση. Τζας, για δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον συντονιστή για την έκθεση αυτή την οποία συνέταξε. σύντομα θα είμαι με δύο ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, Μπορείτε να μας διευκρινίσετε για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές από το 2014 μέχρι το 2020. Κάτι θα μπορούσε να μας πει από τώρα σχετικά με τον προγραμματισμό. Και ακόμη κάτι, δεύτερη ερώτηση όσα απαιτούνται και θα πρέπει να συνοδεύουν τα σχέδια αυτά και έτσι να μας προδιαθέσουν για κάτι το θετικό σε αυτές τις προκήρυξεις για το 2012 και τα επόμενα έτη και ακόμα σχετικά με τα νησιά. Τα νησιά γνωρίζετε ότι έχουν ιδιαίτερα ειδικό χαρακτήρα με διάφορες δυσκολίες και εδώ στα νησιά, σε ορισμένα νησιά, τι γίνεται, αυτές οι προϋποθέσεις άραγε θα υπάρξουν όπως τις αναφέρατε εσείς. Μήπως ε, θα μπορούσαν να ληφθούν ειδικά υπόψη αυτές οι προϋποθέσεις κάπως πιο ελαστικές, περισσότερο προσαρμοσμένες στα ίδια τα χαρακτηριστικά αυτών των νησιών. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, <clears throat> ευχαριστώ για την έκθεσή σας περισσότερο από όλους τους άλλους χρειάζεται να ε, αντιμετωπίσετε τα μεγάλα εμπόδια πρώτον απουσία ε, προτεραιοτήτων των κρατών μερών σχετικά με τα λιμάνια. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα κατάλογο λιμανιών που δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους και επίσης πολλοί μου λέγουν ότι η γραφειοκρατία είναι αυτή η οποία καταρακώνει το σύμπαν. Δηλαδή όταν ένας ιδιώτης φορτωτής ο οποίος δεν συνεργάζεται με ένα μεγάλο Ιταλικό οίκο θέλει να ξεφορτώσει στην Ιταλία δεν έχει καμία πιθανότητα και νομίζω ότι τα εμπόδια αυτά μετατοπίζονται από το βορρά στο νότο αυξανόμενα όσο προχωράμε προς το νότο. Εξού και αναφέρομαι στο θέμα αυτό. Όσον αφορά τις, την αυτιλία μικρών αποστάσεων, το short sea shipping, ε, βλέπετε εξελίξεις, βλέπετε να υπάρξουν ε, ε, πιο ενδιαφέροντες, ενδιαφέρουσες μικρές αποστάσεις ε, για την ναυτιλία. Ε, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δικιά σας αντιμετώπιση. Και το ερώτημά μου είναι πώς μπορείτε να βοηθήσετε κατά τρόπον ώστε να υπάρχει καλύτερη κατάρτιση στόχων από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή όσον αφορά το συνδυασμό με την ενδιοχώρα πρέπει να σκεφτώ και τις εμπορευματικές μεταφορές και να κοιτάξω πόσο θα αποσυμφορήσω το όλο σύστημα. Ο κύριος Κουμουτσάκος για δύο λεπτά. μπράβο, βρε παιδί μου. Πες τα Βέβαια το project είναι πολύ μεγάλο και πάρα πολύ φιλόδοξο, αναφυσβήτητα. Γι' αυτό και άλλωστε γίνεστε δέκτης ενός βομβαρδισμού ερωτήσεων και ελπίζω ότι θα μπορέσετε στο χρόνο που θα έχετε στη διάθεσή σας να απαντήσετε σε ορισμένες από αυτές. Ε, και εγώ θέλω να προσθέσω ορισμένα ερωτήματα. Βλέπω στην έκθεση ότι μια βασική παραδοχή του προγράμματος στηρίζεται στο ότι θα χρησιμοποιούνται όλο και μεγαλύτερα σκάφη, όλο και μεγαλύτερα πλοία, με όλο και μεγαλύτερο και περισσότερο εμπόρευμα. Και αυτό βεβαίως έχει μια επίδραση στην υποδομή των λιμανιών που ε, εντάσσονται στο πρόγραμμα. Και όσον αφορά την υποδοχή και όσον αφορά την στήριξη των πλοίων αυτών, την αποθήκευση κτλ. Ε, Πιστεύετε ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει, δηλαδή των μεγαλύτερων πλοίων με τα μεγαλύτερα εμπορεύματα, θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή και η ναυτιλία υφίσταται τις αρνητικές συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης. Μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τα επόμενα 5-10 χρόνια στη λογική ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπαρκτή τάση μέχρι πριν λίγο. Η υπαρκτή τάση για να χτίζονται τόσο μεγάλα πλοία και θα δημιουργούν τις αντίστοιχες ανάγκες ή αυτή η τάση μπορεί να ανακοπεί. Γιατί ήδη καταγράφεται μια ανακοπή αυτής της τάσης. Τώρα όσον αφορά ε, ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό, βλέπω ότι στο νέο σχεδιασμό θα περάσουμε από τα 300 ε, λιμάνια TNT Class A σε 87 λιμάνια, αυτό που λέμε Core Network. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς προσδιορίζονται αυτά τα 87 λιμάνια, πώς φτάσαμε σε αυτή τη μείωση πώς ορίζονται, από ποιους καθορίζονται και αν βέβαια αυτό λαμβάνει υπόψη εθνικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς για τους λιμένες. Ε, είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, διότι είναι μια πραγματικά σημαντική αλλαγή. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αφορά μόνο τους ναυτικούς ή θα έπρεπε κυρίω να εντοπίζεται στους εργάτες στους λιμένες. Διότι είναι θέμα υποδομών και όχι στους ναυτικούς στα πλοία. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο. Ένα, ένα θα ήθελα. Ένα, ένα. Ένα μόνο. Δεν μπορώ κύριε Κουμουτσάκο, ήδη έχουμε καθυστερήσει και υπήρξε αυστηρός για όλους, οπότε δύο λεπτά και τέρμα. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι ο μιλητής θα μπορείτε να συναντηθεί και έξω. Προγράμματα υποδομών, αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να λάβω το λόγο γιατί το σχέδιο αυτό έχει σημασία και απαιτείται ένα συντονισμός. Αυτές οι θαλάσσιες πλωτές οδοί έχουν μεγάλη σημασία και για την μακρινή αυτή περιοχή περπόντια από την οποία προέρχομαι έχει σημασία. Η θάλασσα για μας είναι ιδιαίτερα λοιπόν σημαντική. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τη γεωστρατηγική διάσταση αυτών των περιφερειών των αποκρισμένων πώς συνδέονται με την εσωτερική αγορά και έτσι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τα θετικά σημεία. Ε, και είναι η Ευρώπη η ευρύτερη περιοχή με 25 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, μακρινές ε, περιοχές ε, υπερπόντιες κλπ. Και ακόμα τι γίνεται με τα καύσιμα για την μεταφορά και την αλλαγή προς το φυσικό αέριο να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο την στρατηγική 2020 και να μειώσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και να είναι αποδοτικότερος ο τομέα, Άρα λοιπόν ε, έχει αυτό σημασία για το ολοσχέδιο. Δεύτερο τώρα, για υπηρεσίες και υποδομές έξυπνες ε, για τη σύνδεση όλων αυτών, την παράκαμψη των ε, εμποδίων. Πρόκειται για μια βάση που έχει να κάνει με Γερμανία, την Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία, περιλαμβάνει αυτά τα κράτη και πολλά στοιχεία σημαντικά για την όλη οργάνωση, για τη βελτίωση αυτών των μεταφορών των θαλάσσιων και επίσης τον ανταγωνισμό και θα μπορούσατε να μας πείτε τι ακριβώς φρονείτε. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση του σχεδίου γενικότερα και ακόμα κάτι τελευταίο. Αυτό το ε, ε, με πολλές εισόδους και πολλούς λιμένες. Τι φρονείτε. Τίκα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για την παρουσίασή σας. Μεταξύ των ε, προγραμμάτων που αναφέρατε υπάρχουν μερικά και πόσα που καλύπτουν τη Μαύρη Θάλασσα. Ε, ξέρω ότι υπήρχαν γραμμές του προπολογισμού ε, για ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων και στην Μεσόγειο και στη Βαλτική και στην Δύση και στην Ανατολή. Δυστυχώς όμως ε, για τη Μαύρη Θάλασσα δεν είχαμε γραμμή του προπολογισμού. Να σας ρωτήσω λοιπόν πόσα από τα ε, σχέδια τα οποία αναφέρατε καλύπτουν τη Μαύρη Θάλασσα και επίσης ποια είναι τα βήματα τα οποία μπορούν να αναλυφθούν έτσι ώστε η ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων στην ε, Μαύρη Θάλασσα να συμπεριληφθεί γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια θάλασσα πάρα πολύ σημαντική για την ενέργεια και την προμήθεια ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, την επόμενη χρονιά θα οργανωθεί στην Κωνσταντζα μια ε, συνάντηση για να συζητήσει τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, ε, Όσο γίνεται πιο γρήγορα να απαντήσετε, αλλά να μην ξεχάσετε να δώσετε απαντήσεις και σε όλους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση. διασύνδεση με τις χερσαίες υποδομές. Αρκετά χρόνια πριν είχαμε πει ότι μία από τις προτεραιότητες θα, πρέπει να είναι η σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμένων, αλλά μερικές φορές αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι θα πρέπει να βελτιωθούν κάπως και οι δρόμοι έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό ας πούμε ισχύει στην Πολωνία, στο Γκτάντσκ ε, γιατί δεν είναι πολύ λειτουργική η σιδηρόδρομη προς το νότο και επομένως μεταξύ Γκτάντσκ και Βαρσοβίας ε, πρέπει να είμαστε πολύ, πρέπει να βελτιωθούν οι χερσαίες υποδομές, οι οδικές υποδομές και υπάρχουν προγράμματα για αυτοκινητοδρόμους ε, που θα πρέπει να γίνουν λειτουργικοί πριν γίνουν ε, λειτουργικοί οι σιδηρόδρομοι. η εκπαίδευση, η κατάρτιση των ε, ανθρωπίνων πόρων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Όταν οποτεδήποτε στηρίζω την κατάρτιση, είναι κατάρτιση για όλους για αυτούς που εργάζονται στις ναυτικές εταιρείες αλλά και σε αυτούς που εργάζονται στις εταιρείες επιμελητίας που ασχολούνται με τα logistics δηλαδή. και ξέρετε ότι υπάρχουν ε, ε, δυσκολίες ε, και όσον αφορά το, την πρόθεση των φορτίων. Υπάρχουν πολλά καινούργια στοιχεία, άρα πρέπει να υπάρξει κατάρτιση. Everybody in order to, to, to have the, the possibility of είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αρθούν όλα τα προσκόμματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους. Ο προϋπολογισμός βεβαίως θα πρέπει να αυξηθεί. Γιατί θέλουμε να υπάρχει η διασύνδεση. Μην λησμονούμε ότι η Ευρώπη ότι περισσότερο από το 80% των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διοχετεύεται μέσω θαλάσσης. Και ε, πλέον έχουμε και εσωτερικές μεταφορές ε, φορτίων μέσω θαλασσίων οδών. Εκομπόνους. Το εκομπόνους έδωσε καλά αποτελέσματα στην Ιταλία. Εγώ υποστηρίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εάν δεν είναι δυνατόν ε, να συμπεριλάβει όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον να καλύψει κάποιες ε, από τις ε, περιφέρειες. Είναι ένα καλό κίνητρο. Είμαι υπέρ του η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία να καθίσουν μαζί ε, για να συνομιλήσουν για το θέμα αυτό, γιατί είναι εύκολα μετρήσιμο. Τα ποσά αναφέρονται σε εξωτερικό κόστος και επομένως είναι σχετικώς, εύκολη, σχετικώς εύκολος ο υπολογισμός τους και είναι εύκολο να μεταφερθούν στους οδηγούς και στις μεταφορικές εταιρείες κτλ. Είναι ένα εύκολο διαχείριστο σύστημα. Ε, μου θέσατε και άλλη μία ερώτηση όσον αφορά τον αντίκτυπο των διαφόρων ε, σχεδίων. Βεβαίως γνωρίζουμε το θέμα του αντικτύπου. Γι' αυτό ακριβώς ε, με απασχολεί πάρα πολύ το είδος του καυσίμου και με απασχολεί επίσης και το θέμα της βελτίωσης των κινητήρων που οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν. βλέπετε ας πούμε τα διάφορα σκάφη στους ε, λιμένες και διαπιστώνεται πολύ συχνά ότι ο κινητήρας τους εξακολουθεί να γυρίζει ε, γιατί πρέπει να εξακολουθήσουν να παράγουν ε, ηλεκτρισμό διότι η παροχή ηλεκτρισμού δεν είναι δυνατή από το ίδιο το λιμάνι, από την υποδομή του λιμανιού Συζητήσαμε λοιπόν με διάφορους ε, λιμένες ε, την ε, δυνατότητα αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου έτσι ώστε να παρέχεται στα σκάφη η ενέργεια τη στιγμή, στη διάρκεια μάλλον του ελιμενισμού τους. Και την δυνατότητα ε, οι κινητήρες να λειτουργούν ε, με διπλά καύσιμα, δηλαδή ε, και με το παραδοσιακό καύσιμο και με υγροποιημένο αέριο στη διάρκεια του ελιμενισμού. Αυτά όλα είναι σημεία τα οποία τα συζητούμε. Και αυτή είναι η απάντησή μου σε αφορά την ερώτησή σας. Παραπονιέστε ότι ο υπερ υπερ-εκπροσωπείται στο σχέδιο αυτό. Αλλά αν τα δείτε λεπτομερία, ειδικά τις τωρινές εξελίξεις, θα διαπιστώσετε ότι ναι, αληθεύει ενδεχομένως ότι αριθμητικά σε αριθμό σχεδίων υπάρχει υπεραναφορά του, του Βορρά, αλλά υπάρχουν ένα σωρό άλλα στοιχεία τα οποία ε, αφορούν τις, ε, ε, τις νότιες χώρες. Έχουμε πολλά καλά σχέδια των οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να διευρυνθούν. Επομένως η απάντηση είναι η εξής. Υπάρχουν μικρά κομμάτια στο βορρά, διασύνδεση με την Δανία, με την Πολωνία, με την Γερμανία όντως, αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ σημαντικά, αν όχι σημαντικότερα, τα οποία λαμβάνουν χώρο στο Νότο. The perspectives, ε, Όσον αφορά τις ε, προοπτικές Ελπίζω ότι στα αριθμητικά στοιχεία τα οποία αναφέρθηκα στην αρχή, ε, τα αριθμητικά στοιχεία μάλλον θα τηρηθούν. Βεβαίως εμείς στηρίζουμε την αύξηση του προϋπολογισμού και το ελπίζουμε αυτό. Και ούτως ή άλλως, κατά την άποψή μου, πρέπει να στηριχτεί ο τομέας αυτός. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, δηλαδή ποιες είναι οι απαιτήσει ή προϋποθέσεις, Πρέπει να σας πω ότι αυτές οι προϋποθέσεις αναφέρονται ρητά ε, ε, στην ε, προκήρυξη και εν πάση περιπτώσει όλες οι προϋποθέσεις αποσαφηνίζονται επίσημα πριν από την προκήρυξη. Uh, Να σας πω λοιπόν ότι πέρσι είχα μια συνάντηση στη Μαδέρα σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές. Ε, και στη Γαλλία ήρθαμε σε επαφή με τους υπεύθυνους υπερποντίων διαμερισμάτων. Είδαμε λοιπόν ότι τα περισσότερα από τα γενικά ε, στοιχεία ανίχνευση των ε, σκαφών, και όλα, όλα αυτά τα οποία γίνονται στην ουσία καλύπτουν τις απαιτήσει των, των λιμένων αυτών, των νησιωτικών περιοχών. Συμφωνώ απολύτως ότι η γραφειοκρατία μπορεί ε, και παίζει αποτρεπτικό ρόλο. Έχω επισκεφτεί πολλά λιμάνια και πρέπει να σας πω ότι το τμήμα των ε, υγειονομικών και φυτοϊγειονομικών ε, και κτηνιατρικών ελέγχων είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι. Ε, τα τελωνία γενικότερα είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, αλλά αυτά που αναφέρω είναι ακόμα περισσότερο. Στο κτηνιατρικό έλεγχο οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, ε, και ε, στο, όσον αφορά τις, τους φυτογενομικούς ελέγχους και εκεί μπορεί να παίξει αποτρεπτικό ρόλο η γραφειοκρατία. Πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τους τρεις αυτούς τομείς, δηλαδή τα, τα τελωνία, κτηνιατρικός έλεγχος και φυτογειονομικός έλεγχος. Αναφερθήκατε στην ε, ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων. Βεβαίως μας ενδιαφέρει ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων. Και... Έχουμε 300 ε, λιμένες ε, που είναι πολύ καλοί όσον αφορά την ακτοπλοεία, όσον αφορά την ναυσιπλοεία μικρών αποστάσεων. και υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι νέοι άξονες ε, του, των ΔΕΒ που έχουν εγκριθεί ξεκινούν και τελειώνουν ε, σε λιμάνια. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Στην Ευρώπη που υπάρχουν 300 μεγάλα ε, λιμάνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινητοποιήσουμε το δυναμικό των ε, λιμένων αυτών. Δεν χρειάζεται και ούτε όλες, ε, όλα τα λιμάνια αυτά μπορούν να γίνουν σημεία μεταλιμενισμού, αλλά μπορούν να είναι σημαντικά λιμάνια τουλάχιστον για διασυνδέσεις ακτοπλοείας και ναυσιπλοείας μικρών αποστάσεων. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του μεγέθους των σκαφών. Έχουμε μια κατάσταση Έχουμε τώρα τον Λεβιάθα, να πούμε, που είναι ένα τεράστιο καράβι πάρα πολλών τόνων, χιλιάδων, τόνων και που βεβαίως ε, δεν είναι δυνατόν ε, να ελιμενιστεί σε όλους τους ε, λιμένες. Δεν έχουν όλα τα λιμάνια τη δυνατότητα για τόσο μεγάλα πλοία. Ας πούμε, ας δούμε τι συμβαίνει στο Ρότερνταμ. Όταν φτάνει ένα τέτοιο μεγάλο καράβι, κινητοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις αποβάθρες, γερανοί, και σημαντικός ε, ε, αριθμός ε, σιδηροδρόμων κτλ. Αλλά αυτός ο αριθμός των σιδηροδρόμων δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να ε, μεγαλώσει και επομένως είναι γεγονός ότι έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να έχουμε μια νέα αντιμετώπιση όσον αφορά ε, την χρήση των λιμανιών. Αναφερθήκατε στον Παναμά. Το νέο κανάλι του Παναμά θα ε, εγγενιαστεί το 2014 και τα μεγάλα φορτηγά πλοία θα μπορούν να περάσουν πλέον από εκεί. Θα υπάρχουν ε, μεγάλα πλοία λοιπόν τα οποία θα περνούν ε, είτε μέσω του Παναμά είτε μέσω του Σουέζ ε, από την Ανατολή. Και αυτό είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα έχω μια συνάντηση στο, με το μυαλό στην, ε, στις Βρυξέλλες εδώ. Είχα ήδη μια συνάντηση στην ε, Γένοβα. Ε, τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ε, λοιπόν, όσον αφορά τώρα το, το θέμα των μάλτι ε, multiple getaways. Ε, προχωράει και αυτό. Τέλος, είναι γεγονός ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι ο μεγάλος απόν. Είναι δύσκολο. Επισκέφθηκα και τη Βάρνα και στην Κωνσταντσα και τον Μπουργάς. Υπάρχει μια σημαντική δέσμευση. Είναι ο Βόσπορος που ο ξέρετε είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή. Έχουμε αναλύσει τις δυνατότητες ε, και τα ενδεχόμενα σιδηροδρομικής διασύνδεσης και διασύνδεση βέβαια με τους αγωγούς αλλά γενικά παραμένει το πρόβλημα του Βοσπόρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεολιβέηρα. τρεις επόμενοι συντονιστές είναι ο κύριος Σαβαρή, ε, ο κύριος Ντεβίνκ ε, και θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές οι οποίοι κάλυφθαν ως τώρα και θα ήθελα ε, να αλλάξουμε θέση, θα αλλάξετε και πρόεδρο αλλά προς την κυρία Τικάου παρακαλώ παραμείνετε στα δύο λεπτά διότι ε, ε, έχουμε και τον ε, Επίτροπο Κάλλας οπότε ο χρόνος είναι περιορισμένος. Παρακαλώ τους άλλους τρεις ομιλητές να έρθουν εδώ για να μπορέσουν να ξεκινήσουν με την κυρία Τικάου στην Προεδρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα με, την, ε, ε, με τους συντονιστές των ΔΕΔ. Τώρα σειρά έχει η παρουσίαση του σχεδίου 22 ο παλιός συνάδελφος κύριος Σαβαρή και μάλιστα παλαιός αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών θα είναι ο συντονιστής. Παρακαλώ πολύ αγαπητοί συντονιστές να μην ξεπεράσετε τον χρόνο σας. 10 λεπτά παρουσίαση στις συντονιστές και 2 λεπτά μονάχα για τους συναδέλφους. Έχετε το λόγο κύριε Σαβαρή, παρακαλώ σεβαστείτε τον χρόνο, καταλαβαίνω, αλλά... Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που όταν έρχομαι εδώ, τους πρώην συναδελφού θα ήθελα να χαιρετήσω. Θα προσπαθήσω, για πιο σύντομα, να σας πω ποιο έχει εργασία το PP22 από τη Δρέστη μέχρι την Αθήνα με εθνικές συνδρομικές οδούς που έχετε εδώ στο χάρτη σας έχετε με κόκκινο, κίτρινο και πράσινο. Με πράσινο τι είναι αυτό που έχει ολοκληρωθεί 3.600 χιλιόμετρα μέσα από 7 κρατημέλη και με κόκκινο ε, αυτό που έχει κάπως καθυστερήσει και το κίτρινο ε, προχωράει και αυτό που είναι με διάστηκτη γραμμή προχωράει και αυτό και πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί. Ρίξτε με ματιά στο χάρτη αυτό λοιπόν. Τι θα δείτε, ότι έχει γίνει πολλή δουλειά, τεράστια δουλειά από τη Δρέστη μέχρι τα Ουγγρικά και Ρουμανικά σύνορα. Η Ρουμανική κυβέρνηση καλά προχωράει σε αυτό τον άξονα από τα σύνορα τα Ουγγρικά Κωνσταντζα. Οι Έλληνες επίσης έχουν προωθήσει την νότια στη δομική τους γραμμή αλλά για οικονομικούς λόγους που γνωρίζετε όλοι και καταλαβαίνετε είναι παραμένουν στάσιμη αυτή τη στιγμή και από το βορρά στο νότο έχουμε πρόβλημα ανάμεσα στα σύνορα τα ουγγρικά και τα ελληνικά σύνορα μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Αυτά τα τμήματα που έχουν ε, πραγματοποιηθεί είναι Βρέστη, Πράγα, Βουδαπέστη, μέχρι το Βουκουρέστη, Γεκοστάντατσα, Θεσσαλονίκη, Δομοκό δηλαδή κοντά-κοντά στα βουλγαρικά σύνορα και μέχρι την Αθήνα και μέχρι το 2015 θα έχουμε το τμήμα του γεφυριού, του μεγάλου γεφυριού, το δεύτερο γεφύρι από πολύ πολύ παλιά για τη διάσχεση του Δούναβη στο Βιντίν Καλαφάτ μέχρι τη Ρουμανία και στην Τσεχία θα πρέπει να ολοκληρωθεί κανονικά ο άξονας Χέντιν με τα γερμανικά σύνορα, τη γερμανικά σύνορα και την Πράγα και ο νότιος ε, άξονας επίσης μέχρι το Λίντς. Στη Ρουμανία κανονικά θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί ο άξονα Μπέκε Σαββάν Κούρτιτσι στα σύνορα και μέχρι το Σιτζοάρα τη Μισοάρα, στην ε, ανατολικά της Ρουμανίας και ελπίζουμε ότι ε, από τη Δομοκό και πάνω θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε όπως και με Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και αυτό το δίκτυο βλέπουμε ότι λειτουργεί ακόμα καλύτερα από τη στιγμή που συνδυάζεται με εθνικές προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε διευρωπαϊκά σχέδια αν ε, δεν τα θεωρούσουν ε, τα κράτη σαν εθνικής προτεραιότητες ε, έχουν μεγάλη σημασία αυτά και έτσι υπάρχει ένα σχέδιο διαχείρισης που να λαμβάνει υπόψη την διάσταση αυτή. Μετά το 2015, για να προχωρήσουμε, έχουμε και την αλίστρια εδώ, δεν θα μακρηγορήσω. Από την Ρεβέργη μέχρι τα τσεχικά σύνορα έχουμε ένα πρόβλημα η Γερμανία δεν θα ήθελα να αναπτύξουν ε, με τα ίδια πρότυπα εκεί γιατί δεν είναι προτεραιότητα γερμανική και θα πρέπει να διοργανώσουν αυτή είναι εθνική τους προτεραιότητα, το εθνικό τους δίκτυο. Δεν είναι ότι δεν θα επανέλθουμε σε αυτό. δεν μας δίνουν από τώρα μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Θέλουμε να το εντάξουν στην επόμενο γερμανικό πρωτα γραμματισμό υποδομών. Και επίση ένα μικρό τμήμα στην Ουγγαρία, Τάτα Βούδα, Πέστη, ένα σύντομο τμήμα, βραχή τμήμα, και κράιοβα Σόφια ε, και τα σύνορα με την Ελλάδα. Το τμήμα αυτό, την κόκκινη αυτή γραμμή που βλέπετε έχει ιδιαίτερα καθυστερήσει, το διαβάσατε και στο έγγραφο. Συμπέρασμα, όταν αποκλίνουν οι εθνικές πατρίδες από τις ευρωπαϊκές, τότε δεν προχωράνε τα πράγματα και αν η γεωγραφική κατάσταση είναι δύσκολη επίσης. Και ακόμα ένα πρόβλημα ε, και ένα παράδειγμα. Το Βιντίν Καλαφάτ, ε, κοιτάξτε το γεφύρι αυτό, πολύ καλό έργο, με μερικούς μήνες καθυστέρηση, κανονικά θα εγκαινιαστεί την επόμενη χρονιά στο PP22 e εντάσσεται ένα γεφύρι που θεωρητικά που εδώ σας παρουσιάστηκε σαν συνδρομικό και οδικό γεφύρι. Ρίξτε μια ματιά τώρα την επόμενη φωτογραφία και με την πρόσβαση τη συνδρομική. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα που θα πρέπει να ρυθμίσουμε στα σύνορα. Πολύ μεγάλα έργα, υπέροχα, αλλά δύσκολη και καθυστερή πρόσβαση συνδρομική. Πρώτα απ' όλα θα εξυπηρετήσει οδικά και επίσης ε, για την διαχείριση αυτή τη μεθοριακή πρέπει να καταβληθεί την προσπάθεια ώστε να περνάνε και τα τρένα μια κάποια μέρα. Και την πρόσβαση τη από Βιντίνα από βουλγαρικής πλευράς αλλά από ρουμανικής πλευράς έχουμε 11 χιλιόμετρα και μέχρι την Γκράγεβα που είναι στα 80 χιλιόμετρα χρειάζεται 4 ώρε. Ε, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το πετύχουμε όταν έχουμε παρόμοια υποδομή. Θα πρέπει και από δύο πλευρέ να χαράσονται και να πραγματοποιούνται οι γραμμέ. Αυτή είναι η διαχείριση η διαμεθοριακή που θα πρέπει να ισχύει. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το πολύ καλό, αλλά δεν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση. Δεν είναι ότι φταίει κάποιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα την ίδια στιγμή. Ο δικό μα ο ρόλο είναι να δώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια ώστε όλα αυτά να προχωρήσουν. Τώρα από πού, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις, στο Νότο κυρίως για να βελτιωθούν τα πράγματα από δική πλευρά στι ανατολικέ χώρε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και σε αυτό ενδιαφέρεται ο πληθυσμό. Επίση, από κοινωνική πλευρά δεν υπάρχει κατάλληλο συντονισμό και ακόμα άλλε μη συντονισμένε με ευρωπαϊκέ προτεραιότητε προσπάθειε. Άρα λοιπόν δεν προωθούνται και ένα πρόβλημα ανάμεσά μας συντονισμού ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τραπέζα και στις ε, διευθύνσεις της περιφερειακή και η Δυσμούβ είναι εκείνη που χαράσει την πολιτική μεταφορών και η περιφερειακή που ε, ε, χρηματοδοτεί, αλλά χρηματοδοτεί άλλες προτεραιότητες. Η πρώτη λέει θέλω τρένα και η δεύτερη που χρηματοδοτεί δρόμους αρκετά σημαντικό σαν πρόβλημα. Προσπαθώ να ρυθμίσω όσο γίνεται ανάμεσα σε αυτές τις χώρες ανατολικά του PP22 e με ένα τμήμα συντονισμού που συνεργαζόμαστε όλοι αυτοί που προανέφερα. Να συνεχίσουμε τώρα. Λόγοι καθυστέρησης. Για κοιτάξτε. Το πράσινο του PP22 είναι ιδιαίτερα δύσκολο γεωγραφικά για τη χάραξη. Και μετά στα κόκκινα βλέπετε τον δρόμο των Βαλκανίων πιο γρήγορος, σε καλύτερη κατάσταση και με ηλεκτροδότηση ευρύτερη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαλέξουμε. Ε, εδώ εμείς ε, οι Ευρωπαίοι επενδύουμε στο πράσινο, αλλά και το, το κόκκινο είναι φυσικός δρόμος, ας το πούμε έτσι. Για τα κράτη-μέλη όπως για Ρουμανία και Βουλγαρία είναι μας πιο δύσκολο να βάλουν εκεί δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα τμήματα που πάνε από τα σύνορα τα ουγγρικά στα ελληνικά σύνορα. Οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι έχουν τις δικές τους ε, φυσικές προτεραιότητες. Είναι από την Ανατολή στη Δύση, για την Κωνσταντζα ας πούμε να καταλήξει, για να βελτιωθεί η ρουμανική οικονομία. Επίσης σημαντικές ε, αστυνομικές μεταφορές προς την ε, κεντρική Ασία. Περισσότερο τους ενδιαφέρει αυτό, αλλά πάνε στα νότια. Ε, στη Βάργκε και στο Μπουργκάς θέλουν να πάνε επίσης οι γειτονές τους. Καταλαβαίνετε εδώ ε, όλα αυτά οι προτεραιότητες ε, βλέπουμε ότι είναι από βορρά σε νότο που κοστίζουν ενώ τα ίδια τα κράτη θέλουν να καταλήξουν στη Μαύρη Θάλασσα αυτή η δρόμη. Βλέπετε λοιπόν, ίσως έχουν και δίκιο στη στρατηγική τους. Για να δούμε λοιπόν τι κάναμε. Πώς θα διαχειρίζονται όλα αυτά ξεχωρίζοντας τα δύο αυτά του PP22. Πρώτα απ' όλα Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία δεν λειτουργεί τόσο καλά εκεί η υποδομή, αλλά έχουν προχωρήσει τα πράγματα περισσότερο και Ουγγαρία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία που δέχτηκαν ε, να έχουμε μια ομάδα πιλότο που να συνεδρίζει ένα εξάμεινο για το πώς έχει κατάσταση την πραγματοποίηση αυτών των έργων και έτσι να μας συνοδεύει και ο Ροδανδιστικός Φορέας η Γενική Move, η Περιφερειακή και η Τράπεζα και έτσι επιτόπου με μια κατάλληλη προσέγγιση από, πάνω προς, από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Κάθε έξι μήνες θα βλέπουμε πώς προχωράνε οι εργασίες και τι γίνεται, ποιες διορθώσεις θα πρέπει να επιφέρουμε. Τον Οκτώβριο συναντηθήκαμε για πρώτη φορά μέσω μιας υπουργικής συμφωνίας της 2 Δεκεμβρίου του 2010. Επίσης δύο μελέτες οι οποίες έχουν ξεκινήσει μία για να έχουμε την ακριβή εικόνα της όλης γραμμής είναι πολύ καλή τα κράτη-μέλη βρήκαν ένα γραφείο μελετών ε, από την Ελλάδα, ελληνική εταιρεία, μας έκανε τα πάντα, μας έδειξε ακριβώς ακόμα και την, ε, την ταινία βλέπουμε εδώ πέρα, τα τρένα που περνούν και βλέπετε αυτά τα παραδείγματα, είναι πολύ καλή δουλειά. Άρα λοιπόν ανάλυση ε, ε, χρόνος, ε, επιχειρησιακή ταχύτητα, όλα αυτά, γεωγραφικά πώς έχουν τα πράγματα και ενδεχόμενες αλλαγές στη γραμμή. Ξεκινώντας από τη μελέτη αυτή, ξεκίνησε μια καινούργια για την κυκλοφορία για τη ροή της κυκλοφορίας Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνουμε σε βάθος ε, στην όλη διαχείριση αλλά και διαμεθοριακά μεταξύ Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Βλέπετε στο καλαφάτε αυτό για να δούμε τις επενδύσεις που θα γίνουν σε αυτό το τμήμα κοντά στα σύνορα και πολλά περιμένουμε από τις ευρωπαϊκές πιστώσεις για, τις για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική όπως θα ψηφιστεί βέβαια η κρίση ε, πάει σε αυτές τις χώρες και η Ελλάδα που δεν ξέρει τι θα κάνει με τον προγραμματισμό των επενδύσεών της. Λιγότερο κάπως η Ρουμανία, αλλά το Διεθνές Νομιστικό Ταμείο ελέγχει εκεί την κατάσταση, βλέπει τα πράγματα, εξετάζει τα πράγματα, θα πρέπει να δούμε και ακόμα κλείνουν γραμμές οι Ρουμάνοι για να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε ορισμένες γραμμές. Δύσκολη λοιπόν η κατάσταση. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες που λειτουργούν καλά και σωστά, είναι ιδιαίτερα δραστήριες από τη στιγμή που μπορεί να κατανοήσει και να προσαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εθνικές προτεραιότητες αλλά και βοηθήσει για να διαχειριστούν τον χώρο του στον εθνικό. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη διαχείριση επιτόπου και όλα αυτά θα βελτιωθούν, θα αναπτυχθούν και θα καταλήξουν σε επίπεδο Βρυξελών. Αυτά ε, μπορώ να σα πω τόσο σύντομα. Σας ευχαριστούμε Ευχαριστούμε κύριε Σαβαρή. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινέσκου. Κυρία... Ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Στο νέο δίκτυο το οποίο θέλει να καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπάρχει διαχωρισμός σε δύο διαδρόμους. Στην ε, <clears throat> Ουγγαρία λοιπόν υπάρχει ε, μία διακοπή διότι το ένα τμήμα ανήκει στον ένα διάδρομο και το άλλο σε άλλο διάδρομο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς εσείς διαβλέπετε την κατάσταση και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός. Δεύτερον, μιλήσατε για χρηματοδότηση. Εις, την ανακοίνωση συνδέοντας την Ευρώπη ελέγχθη ότι η ευρωπαϊκή συμμετοπή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 20% του κόστους του προγράμματος. Τι σημαίνει αυτό. Χρηματοδότηση από το Connecting Europe ε, και από τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, συνολικά δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος, διότι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ χαμηλό αυτό το επίπεδο. <clears throat> Επίσης, ε, ε, όσον αφορά την εξάρτηση της χρηματοδότησης ε, από το Connecting Europe και από την αφομίωση των πόρων στη δημιουργία αυτού του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ε, αντιλαμβάνομαι επιπλέον ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά το κόστος των διαφόρων προγραμμάτων PP22 e και ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, εδαφολογικές ιδιαιτερότητες υπάρχουν μεγάλες μεγάλο κόστος και μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Να ρωτήσω κάτι μετά πως άκουσα πλευράς Μαρινέσκου αυτό το νέο μέσο Connecting Europe και επίσης πως αυτό κατανέμεται σε δύο διαδρόμους στο TEN. να ρωτήσω κάτι. Ε, ο συντονιστής διαμαρτύρεται επειδή δεν υπάρχει ή κατάλληλο συνδυασμό ε, λόγω εθνικών προτεραιοτήτων. Θα ήθελα να καταλάβω κάπως τι γίνεται ανάμεσα Ανατολή και στη Δύση, πώς έχουν αυτές ε, οι συνδέσεις, έχει σημασία για την ε, Δημοκρατία της Τσεχίας, όπως επίσης Γερμανία, Τσεχία ειδικότερα, ανάμεσα στην Πράγα και στην Ιρεμβέργη και ανάμεσα στην Πράγα και στο Μόναχο. Αυτά τα σχέδια έχουν συμπεριληφθεί για την επόμενη περίοδο ανάμεσα στις προτεραιότητες. Θα είναι ρεαλιστικό να σκέφτεται κανείς ότι θα έχει ε, μια κάποια χρηματοδότηση, μάλλον χρηματοδότηση και ακόμα στο σημείο που στη διαδρομή που πάει από την Πράγα προς τα Ανατολικά. Αυτό η χάραξη έχει γίνει στο μεγαλύτερο μέρος της αλλά τι γίνεται, τι φρονείται για τη δυνατότητα να μπορέσει κανείς να ενισχύσει στον Πέρνο, τον κόμβο αυτό. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ, <clears throat> ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την έκθεση. Έχω ορισμένε ερωτήσεις, τις οποίες άλλωστε ε, έχω λάβει από τσέχους συναδέλφους οι οποίοι κοίταξαν ε, το χάρτη του δικτύου και τον χάρτη των ε, διαδρόμων ε, και έχουν ερωτηματικά. Όταν υπάρχει σύνδεση προς τη Βιέννη προβλέπονται δύο αυτοκινητόδρομοι ή τουλάχιστον δύο οδοί σε 50 έως 70 χιλιόμετρα απόσταση και τα δύο είναι στο Core Network. Έχει νόημα γεωγραφικά, διότι γεωγραφικά δεν μπορεί να είναι ε, ε, λογικό αυτό. Γνωρίζω την ε, περιοχή καλά. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας διαχωρισμός διότι εδώ αυτό που μας απασχολεί είναι όταν υπάρχει μία διέλευση των συνόρων μεταξύ Τσεχίας και Αυστρίας όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα με την Natura 2000 αν έχουμε έναν βασικό διάδρομο και κάνουμε δύο συνδέσεις προς το Μπρουν ε, μήπως δεν θα μπορούσε κανείς έτσι να απλοποιήσει διότι ε, δεν μπορεί κανείς ε, να πείσει ότι χρειάζονται δύο ε, αυτοκινητόδρομοι με μικρή απόσταση μεταξύ τους στο κεντρικό δίκτυο. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπέργκερ κύριος Κόχλιτ. Σας ευχαριστώ. Εδώ η διαφορά τώρα αυτό, σε αυτό που συνέβαινε πριν από 8 χρόνια εντάξει μπορώ να να μιλήσω και άλλη γλώσσα επιτέλους ε, στην Πρίσλα και Μπρατισλάβα βλέπουμε το τι συμβαίνει και να συμπληρώσουμε τη σύνδεση με την Ιρεμβέργη από πλευράς της Αιχικής. Αυτό το, αυτή η διαδρομή θα μπορούσαμε να την βελτιώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε διπλή συνδρομική γραμμή, είτε ένα μια διαδρομή υψηλής ταχύτητας. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά αυτή τη διαδρομή ε, αρκετές φορές ε, ε, έχω ταξιδέψει. Επίσης Μπουτιόβιτσα και Λίντς, το κομμάτι αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύντομα. Και γνωρίζω ότι ε, δεν ενδιαφέρονται όλοι στη σύνδεση αυτή για τη σύνδεση αυτή, αλλά χαίρομαι που επιτέλους καταφέραμε να διαπραγματευτούμε το κομμάτι που συνδέει την, τα τσεχικά σύνορα με το μόναχο της Βαβαρίας. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί. Κοχ. Ευχαριστώ τον πρώην συνάδελφό μας κύριο Σαβαρή. Νομίζω ότι ο διάδρομος 22 είναι πολύ βασικός και συνδέει την Ελλάδα με την κεντρική Ευρώπη και έχω τρεις ερωτήσεις. Υπάρχουν βασικές διαφορές όσον αφορά τον προγραμματισμό και την πρόοδο ε, εξελίξεως μεταξύ των χωρών. Σκέφτομαι εδώ τις πρωτοβουλίες των πολιτών στις διάφορες χώρες. Μπορούμε να διδαχτούμε από αυτές, δηλαδή μεταξύ των νοτίων χωρών και της Αυστρίας με τη Γερμανία. Επίσης, όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, υπάρχουν σημεία μεταφορτώσεως για να πάει κανείς από το σιδηρόδρομο στο ποτάμι ε, ή στην ε, οδό και επίσης ποιο είναι το μέλλον αυτών των δικτύων εάν η Ελλάδα δεν υπερβεί την κρίση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα και εγώ να κάνω μία ερώτηση προς τον κύριο Σαβαρή. Ε, στην έκθεσή σας του 2010 είχατε αναφέρει σοβαρά προβλήματα σε την περιοχή και είχατε πει ότι προς ε, την Βράιλα και την Κωνσταντσα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι το 2015 και να έχει χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα. Ενώ στην έκθεσή σας λέτε ότι για διάφορα τμήματα Έχουμε το σύστημα ERTMS το οποίο έχει εφαρμοστεί και θέλω να σας ρωτήσω τι πιστεύετε για την ιδέα της εφαρμογής του ERTMS για ολόκληρο το σύστημα. Το λόγο έχει ο κύριος Σαβαρή. Oui, alors, euh, ναι, να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μαρινέσκου, έχετε δίκιο. Δεν το έχουμε θετήσει ακόμα, το αντίθετο, αλλά έχουμε τις νέες προτάσεις. Είχαμε και ένα χάρτη εδώ, ίσως θα μπορούσε να παραμείνει, γιατί θα μας χρησίμευε. Το PP22 e πάει σε δύο διαδρόμους, σε ένα καφέ από το Ρόστοκ μέχρι το Μπειραιά και ένα καινούριο στοιχείο που ζήτησα και έχει συμπεριληφθεί μέχρι Μπουργκάς και Βάρκα, Βάρκα, που ήταν η προτεραιότητα της Βουλγαρίας μέχρι εκεί να πάει και μετά στο μπλε αυτό το γαλάζιο μάλλον από το Στρασβούργο μέχρι την Κωνσταντζα. Έτσι. Α, λοιπόν το PP22 έχει δύο κλάδους, δύο τμήματα που πάνε μακρύτερα γιατί είχαμε τώρα, έχουμε τώρα τη γραμμή που πάει μέχρι το Ρόστοκ και από την Βέργη μέχρι Στρασβούργο, καταλαβαίνετε. Θα δούμε τώρα τι θα, πώς θα αντιμετωπίσετε τις προτάσεις της Επιτροπής. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί απαντούν στην ερώτηση Γκορ νομίζω που λέει ότι έτσι ε, αυτά τα τμήματα θα μπορούσαν να συνδυαστούν, να ασχοληθούμε με την όλη ανάπτυξη διακομβική, να εργαστούμε και για τον κόμβο και για τις διάμεσες πλατφόρμες, ε, Δούναβη και στη στονομική γραμμή PP22, e πώς θα συνδυαστεί η οδική σύνδεση με τη συνδρομική. Αυτό είναι το πλέον έκτιμα αυτής της πρότασης που είναι σφαιρική, διακομβική και είναι ε, κάτι παραπάνω από σκέτα, θαλάσσια, ποτάμια, οδική κλπ. Άρα λοιπόν ε, προσθέμενη αξία και δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με το καφέ διάδρομο. Ασχοληθώ με το ένα με το άλλο. Θα πρέπει να δω αυτό το πράγμα. Ε, να δούμε πώς θα προχωρήσουν ομιλίες στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά μέχρι το 2013 θα ισχύσει. Παραμένουμε στο PP22. E Εντάξει. Τώρα για το κόστος. Το Connecting Europe Facilities είναι 20% αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και το Ταμείο Συνοχής 80-85% της πίστοσης ε, στην χώρα που συμμετέχει. Το 20% είναι ο περισμός εκεί που δεν ανήκει σε αυτές τις χώρες, αλλά έχουμε πιστώσει πάντα από το Ταμείο Συνοχής και το Connective Facility έχει αυτό το ειδικό, το ειδικό στοιχείο. Η DG, η Γενική Διεύθυνση MOVE, μπορεί να τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει το ύψος των πιστώσεων, γιατί θυμάστε ότι ε, δεν υπήρχαν πολλά χρήματα εκεί, 8 δισεκατομμύρια 3, τώρα θα έχουμε 31,5 δισεκατομμύρια, μια σφαιρική ε, με ένα σφαιρικό ποσό που θα, ε, ακόμα ψηλότερο που θα έχουμε και την ενέργεια κλπ. Αυτά η connecting facility θα ήταν 20% το πολύ στις χώρες από τουρκική πλευράς αλλά εντάξει επαρκούν γιατί σε αυτό το τελευταίο κανονισμό τον δημοσιονομικό πήγαμε στο 25% αλλά ποτέ δεν τον πετυχαίναμε. Έτσι στιγματοδότηση υποδομή στα παλιότερα κράτη-μέλη. Εγώ επί τόπου εργάζομαι και μερικέ φορέ είχαμε 10-15% και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση στο δημοσιονομικό κανονισμό ε, πίστευαν από μια μεριά ότι είχαμε 25, αν είμαστε 5-10, πολλές φορές κάπου εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και πολλές δυσκολίες, αλλά δίκιο έχετε τώρα που αντιμετωπίζουμε αυτή την κρίση για τα κράτη όπως η Βουλγαρία και όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και ακόμα χειρότερα στην Ελλάδα ούτε 20% καλά-καλά δεν μπορούν να συνεισφέρουν και αυτό μας δημιουργεί μια κάποια ανησυχία. Κυρία μου, για το τμήμα ανάμεσα στην Γερμανία και στην Τσεχία, α, πρόβλημα εκεί. Πολύ λιγότερο τα ανατολικά. Οι Τσέχοι κάνουν τη δουλειά. Σε δύο τμήματα που ξεκινούν από την Πράγα το ένα μέχρι τα σύνορα στη Δρέσδη και στο Σέντιν το άλλο κομμάτι. Στα τσεχικά έχουμε ένα άλλο τμήμα, δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομά του. Τέλος πάντων, και πάει μέχρι την Ιρεμβέργη. Δύο σύντομα τμήματα, Νιρεμβέργη, Σέντιν και Δρέστη μέχρι τα τσεχικά σύνορα. Από γερμανικής πλευράς λοιπόν και εκεί οι Γερμανοί λένε α, καμία προτεραιότητα για να το πραγματοποιήσω. Δεν είναι λοιπόν η προτεραιότητά μου, άρα λοιπόν εδώ παραμένω χωρίς να προχωρήσω. Δεν λένε καμιά φορά εντάξει θα έχουμε τρένα υψηλής ταχύτητας, συντάσσονται μελέτες και αυτό θα γίνει σε 30 χρόνια. Να λοιπόν γιατί δεν κάνουμε κάτι σήμερα. Αλλά αυτό δεν μας ικανοποιεί και ιδιαίτερα. Εγώ προσπαθώ και μάλιστα με ιδιαίτερες δυσκολίες το ίδιο, την διαχείριση, διαχείριση ε, σε Αυστρία, Γερμανία και Τσεχία, σε τρεις χώρες, σε αυτό το τμήμα PP22 για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά σας το λέω ότι υπάρχει μια αντίσταση σαφής, όχι έτσι κρυφή και υπουλή. Μας λέει η κυβέρνηση, ε, μας λέει η κυβέρνηση ότι είναι η προτεραιότητά μου να δω πώς θα βελτιώσω το σύνολο του δικτύου και μια προτεραιότητα από βορρά προς νότο, Augsburg, και πέρα από τα μικρά τμήματα που πάνε Τσεχία. Ε, Βερλίνο-Αουξμπουργκ, απευθεία σύνδεση. Εντάξει, θα το πετύχουμε, πιστεύω, αλλά χρειάζεται διπλωματία, πολύ και άντε πολλά πήγαινε έλα μέχρι το Βερολίνο και στις τσεχικές αρχές πρότεινα μια ομάδα εργασία να προχωρήσει στη Σασίτη στην Πράγα με τους Γερμανούς που εντάξει τουλάχιστον δέχτηκαν να πάνε εκεί για να εργαστούν σε αυτό το σύντομο τμήμα. Αλλά η Γερμανία λέει σαφώς ε, η προτεραιότητά μου είναι η αναδιοργάνωση του δικτύου μου, αύξηση των ε, δυνατοτήτων της και όχι αυτά τα σύντομα τμήματα Άρα λοιπόν και ξεφεύγουν κάπως το παρακάμπτουν λέγοντας, μιλώντας για τα τρένα υψηλής Ναι, απάντησα έτσι. Και μετά Λίντς ε, σύνδεσή του και στο τμήμα αυτό πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό αλλά δεν είναι τόσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τσεχική, Αυστριακή τι λένε. Παλά τα πάει. Εντάξει, μπορεί να μεταφέρει και εμπορεύματα, πάει με 70 χιλιόμετρα την ώρα, δεν θα κάνουμε τώρα τεράστιες επενδύσεις στο για να πάει με 140 χιλιόμετρα την ώρα, να διπλασιάσουμε την ταχύτητα και νομίζω ότι δίκιο έχουν, δεν χρειάζεται να έχουμε ένα αυτοκινητόδρομο ψηλής ταχύτητας. Και από τη τσεχικής πλευράς ποια είναι η προτεραιότητα να έχουν ε, σύντομα οδικά τμήματα στα βράχια και οι Τσέχοι μας λένε εντάξει συμφωνούμε για τη γραμμή αλλά έχουμε πολύ τουρισμό και είναι υπέροχα τα χωριά μας ε, εντάξει αλήθεια αυτό. Πηγαίνετε, επισκεφτείτε τα, όμορφα είναι και θέλουμε να τα προστατεύσουμε τα χωριά μας όπως κάνετε στη Γαλλία μέσω ε, ε, περιφερειακούς ε, γύρω-γύρω από τα χωριά μας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το αδιάφορο από τη στιγμή που ξέρουμε στα χωριά αυτά είναι πραγματικά όμορφα και πρέπει να προστατευτούν. λοιπόν περιφερειακή δρόμη σε αυτούς, αυτή είναι προτεραιότητα. Και αυτό λοιπόν ε, για τους διαδρόμους, ε, για το διακομβικό στοιχείο. Και τώρα για την Ελλάδα έβαλε το RTMS, ε, αλλά όταν φτάνουμε στα ελληνικά σύνορα και τα βουλγαρικά σύνορα, δεν υπάρχει πια τρένο στη Βουλγαρία. Δεν πάει. Δεν δέχεται επιβάτες. Πάει με εμπορεύματα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, τις διάφορες δυσκολίες που παρουσιάζονται και σας το είπα και νωρίτερα ότι αυτός ο δρόμος των Βαλκανίων βλέπουμε ότι για τους Έλληνες έχει σημασία γιατί βγαίνουν από αυτά τα στενά όρια και συνδέονται με το κεντρικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Η κυρία Τικάου τώρα, Κωνσταντσα, πολύ ενθουσιασμός Πολύ καλά τα πάει. Και η ρουμανική κυβέρνηση το θέτει σαν πρώτη προτεραιότητα. Δυσκολεύομαι να πάω προς τα νότια, αλλά για να πάνε προς τα ανατολικά, ναι, εκεί πραγματικά κινητοποιείται ιδιαίτερα η ρουμανική κυβέρνηση και υπάρχουν και κονδύλια που πάνε προ τα εκεί και ορισμένα τμήματα που θα πρέπει να συμπληρωθούν κάπω μπερδεμένα. Είναι δύσκολα, είναι σε ορεινές περιοχές, σε μέσο ύψους όρη και βουνά. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε αυτό τον άξονα με την προτεραιότητα από τα Ουγγρικά σύνορα μέχρι την Κωνσταντσα. Και άντε από εδώ και εκεί κάτι μικρά σύνορα να το την Καλαφάτ, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλή δουλειά, αλλά κάπως περιορισμένο. Περιορισμένη είναι γιατί είναι ε, σε αυτόν τον άλλο άξονα. Αυτά λοιπόν, ε, ε, αυτά θα σας πω, ελπίζω να κρυβολόγησα. Σας ευχαριστούμε κύριε Σαβάρη, λέει πρόεδρος, κύριε Τικάου. Οι συνάδελφοι με συγχωρείτε, <clears throat> είχα ζητήσει και εγώ το λόγο και δεν μου το δώσατε. Μπορώ να πω κάτι. Καταρχήν για το, την Ιρεβέργη ΚΕΠ είναι ένα θέμα αλλά ό,τι δεν ενδιαφέρει τους σιδηροδρόμους δεν ενδιαφέρει τους Γερμανούς εκτός από τη Βαβαρία. Γι' αυτό με την Πολωνία από το 1972 είχαμε όπου είχαμε 18 συνδέσεις, τώρα έχουμε μόνο 10 και χωρίς πλήρη ηλεκτρική σύνδεση. Η κατάσταση αυτή στη Γερμανία είναι τραγική μετά όσον αφορά την γέφυρα είχαμε πει ότι στο Δούναβι σε μία απόσταση 100 χιλιόμετρων δεν υπάρχει δυνατότητα να διέλθουν αυτοκίνητα ή πεζοί και χρειάζεται μία γέφυρα. Μετά, Πράγα, Βίνη. Ε, υπάρχει δυνατότητα συνδέσεως μέσω του Λίντς και του Μπρούνεν. Ε, μήπως ε, ξέρουμε τι γίνεται για τον πριν ενδιαφέρεται η Τσεχία αλλά θα γίνει ένα σιδηροδρομικός σταθμός ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση και γι' αυτό ενδιαφέρει τους Τσέχους. Αλλά αν δεν πάρει χρήματα όπως δεν πήρε και η Στουτγάρδη, μήπως μπορούν να ξέρουμε τι μέλη να γίνει από όλα αυτά. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω σε όσα βρίσκονται στο PP22, δεν το γνωρίζω. Τα υπόλοιπα τα ξέρω όμως ε, Αυτό το πρώτο. Και μου ζήτησατε πέρυσι, ναι, το συνέχισα. Προσπαθώ να έχω βίντεο καλαφάτ, να έχω και ένα διάδρομο, μια λωρίδα για τα ποδήλατα. Ε, εντάξει. Ε, ναι, μου έχουν πει, αλλά θα τα δούμε όμως σίγουρα τη μέρα που θα γίνουν τα εγγένεια. Εντάξει, πάντως αυτά που ζητάτε εγώ τα προώθησα και ακόμα μελέτες σχετικά με κυκλοφορία κάνουμε για να δούμε τι γίνεται. Γιατί όταν υπάρχουν περισσότεροι ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σόφια με τρένο και ότι το τμήμα αυτό είναι, στοιχίζει πολλά δισεκατομμύρια. Πρέπει να δούμε τον αριθμό των επιβατών και αν είναι μεριά τόσο υψηλό κόστας. Ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχίσουμε. Η Γενική Διευθυνσή μου λέει εντάξει Ίσως ε, θα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικό τρόπο. Με συγχωρείτε σύντομα σύντομα, δεν ξέρω αν ε, σας κάλυψα πλήρω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σαβαρίλη, λέει Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε πολύ πίσω στον ε, προγραμματισμό μας και στη μερίχια διάταξη. Ο Επίτροπος Κάλας τελικά θα έρθει το μεσημέρι της 20 Δεκεμβρίου και όχι σήμερα. Γιατί δεν θα έχουμε τελειώσει. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω από τον κύριο Κάρελ Βίνκ, ο οποίος είναι συντονιστής του ERTMS, να, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα είμαι λίγο πιο τεχνικός εγώ σε σχέση με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες αδελφή μου ε, γιατί είναι οριζόντια, είναι ε, κάθετα μάλλον υπεύθυνοι για τα θέματα τους, ενώ εγώ είμαι οριζόντια. Θα σας μιλήσω για το σύστημα ERTMS και αυτό που θέλουμε είναι να μεταφέρουμε, να μετατοπίσουμε την μεταφορά εμπορευμάτων στον σιδηρόδρομο μέσω δύο τρόπων. Πρώτον, μέσω της ε, διαλειτουργικότητας και της χρήσης των ε, προαναφερθέντων διαδρόμων. Όταν αρχικά σκεφτήκαμε την εφαρμογή αυτού του συστήματος ERTMS, ε, είχαμε ενσωματώσει έξι ERTMS διαδρόμους, αλλά η ιδέα και η δικιά μας και του Επιτρόπου είναι να γίνει πιο συνεκτική η αναφορά των διαδρόμων, γιατί υπάρχει σύγχυση όσον αφορά το θέμα αυτό και επομένως αυτά που θα σας πω ισχύουν για όλους τους διαδρόμους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι εξ αρχής. Ε, ε, όταν ασχολούμαστε με τεχνικά προβλήματα όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε το θέμα ε, των οικονομικών λόγω της κρίσης και των οικονομικών δυσχεριών. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω κάτι που έχω ήδη ξαναπεί ενώπιόν σας. Δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν από οικονομική άποψη να αιτιολογήσει κανείς το ERTMS. Μπορεί όμως να δικαιολογήσει άλλα, τρία άλλα πράγματα ε, όσον αφορά τους διαδρόμους που συμμετέχουν στο ERTMS. Πρώτον, να αρθούν τα προσκόμματα, δεύτερον να χρησιμοποιηθεί το ERTMS και τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και θα επανέλθω σε αυτό, ε, η πιστοποίηση οι κανόνες πιστοποίησης, συμμόρφωσης. Εξ αρχής είπαμε, όταν ξεκινήσε η δουλειά ε, με την ε, ε, Κομισιόν, είπαμε ότι θέλουμε χρειαζόμαστε απαραίτητα ενιαία πρότυπα, ενιαία στάνταρ την Ευρώπη και μέσω μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει το 2008 πρώτον θεσμοθετήσαμε το πρόγραμμα το οποίο ισχύει σήμερα και στο ίδιο μνημόνιο κατανόησης αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα που θα βασίζεται στο σύστημα 000 ακριβώς ε, γιατί μπορούμε ε, εκ των υστέρων να προσθέσουμε λοιπές διαλειτουργικότητες η γραμμή 3, η γραμμή βάσης 3 που θα προχωρήσει το 2012 με ε, πραγματική θέση σε ισχύ το, 2015 ε, θα είναι προσαρμοσμένη ε, στα, στο 000D. Γιατί λέμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί το ERTMS, γιατί ακούμε πάρα πολλές επικρίσεις για το σύστημα, αλλά πρέπει να επαναλάβω ότι προοδεύουμε. Σε 14 χώρες μέλη έχουμε 7.000 χιλιόμετρα που ε, ε, ε, έχει υλοποιηθεί το ERTMS. Επίσης, αρκετές χώρες μέλη αποφάσισαν ε, να μεταφέρουν ε, ολοκληρωτικά το σύστημά τους σε ERTMS, είτε γιατί το σύστημα ήταν παπαλαιωμένο, είτε για λόγους ασφαλείας. Αλλά το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Αυστρία, οι κάτω χώρες, το Βέλγιο, καθώς επίσης και η Ελβετία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ολοκληρωτικά να μεταφέρουν το σύστημά τους σε ERTMS. Επομένως, προφανώς κάποια πλέον εκτήματα πρέπει να υπάρχουν. Αυτό που επήγει τώρα είναι ότι μέχρι τώρα είδαμε το ERTMS σε εθνικό επίπεδο, αλλά περνάμε τα σύνορα ε, και επομένως εδώ ε, υπάρχει δυσκολία στην διέλευση των, των συνόρων έστω και αν έχουν γίνει πολλές ε, ε, πρόοδοι μεταξύ του Περπινιά και του Φιγκέιρας στην, ε, μεταξύ δηλαδή Ισπανίας και Γαλλίας έχουν γίνει πάρα πολλές πρόοδοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το σύστημα αυτό πρέπει να στεφθεί από επιτυχία. Και ένα τέταρτο πράγμα θα ήθελα να υπογραμμίσω σχετικά με το ERTMS και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, σαν Ευρωπαίοι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή είναι αναγνωρισμένο παγκόσμια ε, δηλαδή έχει μεταφερθεί η τεχνολογία. Ε, περισσότερες από 50.000 χιλιόμετρα έχουν ε, δημοπρατηθεί μέσω, για να καλυφθούν από το ERTMS και στην ουσία αν εμείς δεν το εφαρμόσουμε τότε θα χάσει αξιοπιστία το σύστημά μας. Και φαντάζομαι ε, ότι διάφοροι τουλάχιστον από την Ασία θα το βελτιώσουν και θα το εφαρμόσουν οι ίδιοι στις χώρες τους. Αυτά είναι τα επιτεύγματα λοιπόν. Οι δυσκολίες ε, που έχουμε στην, ε, στις φάσεις εφαρμογής ε, είναι πολλαπλά. Πρώτον και για ιστορικούς λόγους ε, οι σιδηρόδρομοι δεν ήταν υπέρ της διατροπικότητας και της διαλειτουργικότητας. Δηλαδή πάντα πολιτισμικά είχαν αυτόν τον περιορισμό. Από τεχνικής απόψεως τώρα έχουμε επίσης το πρόβλημα ότι σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση της ε, υποδομής ε, απαιτεί προσαρμογή σε τοπικές ε, ιδιαιτερότητες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες αιτήσει τροποποίησης είχαμε σε επίπεδο ευρωπαϊκών χωρών. Τρίτον, η διαδικασία συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες συμμόρφωσης εκπονούνται από τις εθνικές ε, αρχές και δεν αφορά μονάχα ε, τις ε, γραμμές και τα λοιπά. Η ελάχιστη αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει το σύστημα, τότε θα πρέπει να ξαναέχετε νέο γύρο για νέες αδειοδοτήσεις από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Και αυτό κοστίζει χώρο, χρόνο και πάρα πολύ χρήμα. Δεν μιλάω για εκατομμύρια, μιλάω για δεκάδες εκατομμύρια. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι δεν έχουμε ακόμα οργανωθεί όσον αφορά την ε, συμμόρφωση στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα επίγον ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Άλλη μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι προμηθευτές προμηθεύουν το, τον εξοπλισμό αλλά ο εξοπλισμός που έρχεται από διάφορες, διάφορους ε, προμηθευτές ε, παρουσιάζει διαφορές. Καμιά φορά ακόμα και ακόμα και για τον εξοπλισμό λύνουμε το ζήτημα, αλλά όταν μιλάμε για, ε, ε, για υποδομή που ε, παρέχεται από έναν προμηθευτή και εξοπλισμό που παρέχεται από άλλον, τότε έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα. Και όσον αφορά τους διαδρόμους. Βεβαίως θα πρέπει να διασφαλιστούν οι επενδύσεις στους διαφόρους, στα διάφορα τμήματα των διαδρόμων έτσι ώστε ε, να προχωρούμε χωρίς δέσμευση. Δεν έχει έννοια δηλαδή σε ένα κράτος μέλος ε, να έχει κανείς ε, άλλα μεγέθη από τη στη διπλανή γειτονική χώρα. Θα ήθελα να επιστήσω την ε, προσοχή όλων για μια ειδική κατάσταση που υπάρχει στη Γερμανία. Η Γερμανία δεσμεύτηκε, οι Γερμανοί είπαν ότι θέλουν να σεβαστούν το ERTMS, αλλά στην ουσία ε, θα ε, εφαρμοστεί βάσει της παλαιότητος του υπάρχοντος συνδρομικού υλικού. Αυτό έχει σαν συνέπεια ε, την ε, γενική καθυστέρηση της ε, Γερμανίας όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των διαδρόμων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι Στη Γερμανία αναφέρεται ότι θα χρειαστούν 4,5 δις για να εφαρμοστεί το ERTMS στο δίκτυό τους. Δεν είναι αληθές αυτό και επίσης το σύστημα STM ε, που δίνει την δυνατότητα ε, σε ξένους ε, να λειτουργήσουν στο γερμανικό σύστημα και ήδη πληρώνουμε γι' αυτό. Πάντως δεν έχουμε δέσμευση της Γερμανίας στο EDP και η στάση της Γερμανίας μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση και σε άλλες χώρες για οι οποίες μπορούν και αυτές να πάρουν την ίδια απόφαση και επομένως ε, τα μεγάλα προβλήματα συμμόρφωσης ε, τα οποία οδηγούν και σε μεγάλα προβλήματα κόστους ε, είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι σε αυτούς και λέω υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε με τη Γερμανία έτσι ώστε να βρούμε ε, μια λύση από κοινού που να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα καλύτερα από ότι ε, την παρούσα συνθήκη. Δεν θα πω τίποτα άλλο για τους ε, διαδρόμους. Νομίζω ότι όλα έχουν αναφερθεί ενδελεχώς από τους συναδέλφους. Προτεραιότητά μου σαν συντονιστού είναι ε, να λειτουργήσει πλήρως το ERTMS έτσι ώστε η βασική γραμμή κιόλας να νομοποιηθεί το 2013 έτσι ώστε να έχουμε πλήρη διαλειτουργικότητα για το 2015 ε, να υπάρχουν κοινά πρότυπα, κοινά στάνταρ για τη διαλειτουργικότητα και το θέμα της συμμόρφωσης να το αντιμετωπίσουμε ε, και βεβαίως να πούμε ότι το ε, ERTMS θα πρέπει να συνδυαστεί με τις επενδύσεις των διαδρόμων. Τέλος, να εξευρεθεί ισορροπημένος φάκελος χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το ζήτημα αυτό πολλοί, πολλές χώρες κοιτούν, βλέπουν το ERTMS σαν ένα επιπλέον κόστος, ενώ είναι βελτίωση, εξυγχρονισμός ε, για το μακροπρόθεσμο ε, μέλλον. 500 εκατομμύρια, ε, επί των οποίων προσθέθηκαν άλλα 100, 600 εκατομμύρια λοιπόν. Νομίζω ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά και θα πρέπει να υπάρχει και η κατέλληλη κινητροδότηση να δούμε λίγο το θέμα των ε, δασμών πρόσβασης ε, ε, στο σύστημα κτλ. Να εξευρεθεί, εν πάση περιπτώσει, η σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες αφενός και τη χρηματοδότηση αφετέρου. Εν συμπεράσματι, θα ήθελα να πω ότι, σαν συντονιστή, αυτό που θα ήθελα να κάνω και σε αυτό στο οποίο θα αφιερώσω τις προσπάθειές μου είναι να υπάρχει καλή και χωρίς πρόβλημα ε, μετανάστευση από τα ισχύοντα συστήματα στο ERTMS. Ε, ε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ασχοληθούν ομού για το ζήτημα αυτό. Δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η μεγάλη προτεραιότητα. μετανάστευση, μεταβίβαση, μετάβαση συγγνώμη, από το ισχύον σύστημα στο ERTMS. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πέντε συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρός πρώτα εν ονόματι του ΕΛΚ. Κύριε συντονιστή, γνωρίζουμε πόσο δεσμευμένος είσαστε για το θέμα αυτό και πόσο τεχνικά δύσκολο είναι το θέμα αυτό και για μας τους ευρωβουλευτές είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε τις τεχνικές δηλώσεις των εμπειρογνωμόνων των διαφόρων χωρών και να επιλέξουμε τη σωστή κατεύθυνση γιατί ξέρουμε ότι είναι βασικά θέματα από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουμε προβλήματα τιμών ή τεχνικών τεχνολογικών προσαρμογών ή ε, και νέα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες χώρες και τα οποία θεωρούνται πλήρως λειτουργικά ενώ άλλοι θεωρούν ότι δεν είναι τόσο προχωρημένα. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ξέρω τι μας προτείνεται για να μην πέσουμε σε μια παγίδα διότι σε ε, πολλές χώρες έχουν γίνει πολλοί περιορισμοί και μία χώρα με αυτό το δίκτυο θα έπρεπε ενδεχομένω να πιστεί πρώτα για να προσχωρήσει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες περισσότερο από ό,τι το έχει πράξει μέχρι τώρα. Ισχύει η πληροφορία ότι με το σύστημα το οποίο επιζητεί η Γερμανία τα σιδηροδρομικά οχήματα των άλλων χωρών θα πρέπει ε, να ε, προσαρμοστούν τεχνικά και ότι τεχνικά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα χωρίς προσαρμογές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η, ε, η λειτουργία στα διά, στις διάφορες χώρες δεν είναι δεδομένη. Επίσης έχει λεχθεί ότι το ποσό το 5 δις δεν αντιπροσωπεύει όλες τις επενδύσεις, είναι και πολλά άλλα μέσα. Ε, ακούμε όμως από πολλές χώρες πόσο υψηλή είναι η δημοσιονομική δαπάνη Τρίτον, όσον αφορά τις επενδύσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα όπως τα βλέπει τώρα η Ευρώπη, εσείς τα θεωρείτε σοβαρά, πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσει, ε, ε, ότι η δέσμευση αυτή είναι δηλαδή μια θετική εξέλιξη. Και τέλος μέσα στα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα θεωρείται ότι το πρόγραμμα αυτό, το σύστημα αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί άμεσα ασχέτως από το νέο συνδέσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Γκρός για να μπορέσουμε να σεβαστούμε την ημερήσια διάταξη και να ακούσουμε και τον επόμενο συντονιστή και να κάνουμε και μερικά ερωτήματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σεβαστείτε το χρόνο σας. Ο κύριος Αλκαντράουι. Ευχαριστώ. Ναι. Θα ήθελα να πω ξεκινώντας ότι είναι σημαντικότατο να έχουμε μια έναν κλωμένο τρόπο αντιμετώπισης ώστε να αντιμετωπίσει ο σιδηρόδρομος την ανταγωνισμό της οδικής σύνδεσης και από τεχνικής πλευράς θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να δω κάνα δυο πραγματάκια που εν μέρη έθεξαν οι συνάδελφοι. Στην παρουσίασή σας είπατε ότι από ό,τι φαίνεται δημιουργούνται νέα εμπόδια. Στις χώρες ε, όπου έχουμε τα δίκτυα MS, ε, τα ειδικέ γραμμές ε, που χρειάζονται τροπολογίες και τροποποιήσεις και προσαρμογές, είτε άλλες αλλαγές που απαιτούνται ακριβώς για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε το συνδυασμό με τα δίκτυα ITMS. Τώρα εσείς σαν συντονιστής τι σκέφτεστε, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτός ο συνδυασμός, αυτή η συνεργασία να είναι δυνατά. Ίσως θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ειδικοί στην... όσον αφορά το θέμα των ε, προδιαγραφών ε, των απαιτήσεων από τα κράτη-μέλη. Και μετά η Γερμανία. Διάβασα εδώ στην έκθεσή σας ότι θέλουν να αναπτύξουν το δικό τους το σύστημα που να συνδυάζεται με το ITMS, αλλά πολλά κράτη-μέλη όπως και η Ελβετία άλλωστε έχουν ιδιαίτερα επενδύσει και ε, εάν η Γερμανία οθετήσει διαφορετικό σύστημα τότε δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει το όλο σύστημα. Και ακόμα τώρα να δούμε μήπως ορισμένοι ε, ανταγωνιστές ε, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν για να προσαρμοστούν σε αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, δεν είναι το καλό το σύστημα. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να πείσουμε τη Γερμανία ώστε να αλλάξει γνώμη και μιλήσαμε για διάφορους διαδρόμους. Ε, αλλά θα πρέπει να δούμε αν όλοι αυτοί θα μπορέσουν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, αλλά έχω δύο τεχνικά ερωτήματα. Ήμουν εισηγητής προ ετών για τα ATMS και τότε είχα πει ότι δεν πρέπει να λεχθεί ότι από τα 20 συστήματα σημάνσεως θα μεταφερθούμε σε 20 νέα διαφορετικά συστήματα για τα TMS. Όταν λοιπόν αποφασίζει κανείς πρέπει να ξέρει κανείς ποιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για να καταρτήσει την, ε, τον διαγωνισμό. Επίσης άκουσα ότι ε, εμποδίζουν τα κινητά, τα, τα κινητά τηλέφωνα την ηλεκτροδότηση των σιδηροδρόμων και επειδή αυτά τα ε, μέσα θα χρησιμοποιηθούν για ε, μία γραμμή από το Βερολίνο προς τη Βαβαρία πιστεύετε ότι θα βλαπτεί από, αυτές τα κύματα των κινητών τηλεφώνων. Επίσης ελέγχθη ότι ε, θα πρέπει ε, οι, ε, ατμομηχανές, οι μηχανές των σιδηροδρόμων αυτών να μπορέσουν να λειτουργούν όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη και ποιος θα τα πληρώσει διότι στην αρχή λέγαμε ότι για τα προγράμματα θα υπήρχε ολοκλήρωση το 2015, τώρα μιλάμε για το 18. Μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία παραβίασης των συμπεφωνημένων και προσαγωγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τι θα γίνει λοιπόν εάν δεν γίνονται σεβαστά ε, τα συμβόλαια τα οποία έχει υπογράψει και η Γερμανία. Τέλος, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά προσόντα ε, ε, ε, εάν πρέπει να πληρωθεί το 80% από το κράτος. Ευχαριστώ η Γερμανία πάντοτε έχει πολλές απαιτήσει και μετά δεν σέβονται τις συμφωνίες. Έχουμε την ε, ευκαιρία να καταρτήσουμε σαφές προδιαγραφές και διαδικασίες κατά τρόπον ώστε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό που αναφέρατε, λέει ο κύριος Κόλιτσεκ, δηλαδή ε, διάφορους προμηθευτές οι οποίοι ε, θα μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνούν. Ευχαριστώ και τώρα δίνω τον λόγο στον κύριο Βίνκ για να απαντήσει. Κύριε Βίνκ έχετε τον λόγο για ε, δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς δεν ακούμε. Uh, θα προσπαθήσω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις και να απαντήσω. Όσο αναφορά την αποδοχή της γερμανικής προτάσεως, χρειάζονται ορισμένες αλλαγές και αν γίνουν αυτές οι αλλαγές θα χρειαστούν νέες διαδικασίες και αν έχουμε να κάνουμε με πολλές χώρες θα χρειαστεί κάποια συμμόρφωση και προσαρμογή η οποία είναι μεγάλο θέμα και οι Γερμανοί μας λέγουν εμείς θα καλύψουμε όλο το κόστος χωρίς όμως να μας έχουν πει ποιο είναι το κόστος αυτό χωρίς να το έχουμε συζητήσει λεπτομερώς οπότε το θέμα είναι ακόμη υποσυζήτηση και ελπίζω ότι στο τέλος οι Γερμανοί θα δεχτούν και άλλες λύσεις. Δεύτερον, αναφερθήκαμε στα 4,5 δις των επενδύσεων είναι η συνολική επένδυση η οποία χρειάζεται όχι μόνο για το ERTMS αλλά και όλων των συνδέσεων στους τέσσερις διαδρόμους που περνούν από τη Γερμανία. Μπορείτε να εφαρμόσετε το ERTMS στις γραμμές που υπάρχουν με τις συνδέσεις που υπάρχουν αλλά θα είναι ανεπαρκής η εποπτεία. Υπάρχουν και μεικτά συστήματα τα οποία έχουμε προτείνει για ορισμό ορισμένους διαδρόμους όπου ορισμένα θα είναι στο RTMS δεύτερο επίπεδο και άλλα με τους παλιούς συνδέσμους αλλά θα διατηρηθεί το σύστημα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες παρανοήσεις και δεν ε, ε, γνωρίζει κανείς ε, τι θα κοστεί το e ERTMS. Θα κοστεί στο 15% μόνο του συνολικού ποσό για όλους τους διαδρόμους. Και βέβαια η υποχρέωση αποτελεί μια δυσκολία γιατί έχετε τα συμφέροντα των κρατών μελών, των σιδηροδρομικών εταιριών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θέλει να τα ενοποιήσει όλα και δεν ε, μπορούμε ε, να δώσουμε ε, κίνητρα βάση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλωστε δεν βλέπω πώς από πλευράς νομικής αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο θέλουν όσον αφορά τα συστήματα. Άκουσα όμως και πολλές ερωτήσεις για τα συστήματα. Η Γερμανία θέλει να αναπτύξει το δικό της σύστημα. Δεν είναι σωστό αυτό, διότι όπως σας είπαμε η Γερμανία θέλει να εφαρμόσει το ERTMS. Δεν το ξανααμφισβητούμε. Θέλουμε να φτάσουμε στο επίπεδο 3. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά η Γερμανία προς το παρόν δεν είναι έτοιμη να εξοπλίσει τους διαδρόμους και ιδίως τις δεσμεύσεις που υπάρχουν για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και έτσι είναι μπλοκαρισμένοι και επανέρχομαι τώρα σε ένα θέμα όπου ελέγχθη ότι τι θα κάνουν οι γειτονικέ χώρες, η Ελβετία, η Αυστρία, η ε, Ολλανδία. Εχθές ε, παρέστην σε μία τέτοια συζήτηση όπου υπήρχαν και οι τέσσερις εταίροι του διαδρόμου Ρότερνταμ Τζένοβα και μου εξήγησαν ότι για αυτούς το ETM που προτείνει τώρα η Γερμανία είναι ανέφικτο, πολύ δαπανηρό, δεν λύνει το πρόβλημα και καθυστερεί τις ε, επενδύσεις και δεν αντιλαμβάνονται γιατί πρέπει αυτοί να καθυστερήσουν τις επενδύσεις τους λόγω των Γερμανών. Το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι δύσκολο και το μόνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι πρέπει να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση για τις διάφορες προπτικές. Ζητήθηκε από τη Γερμανία να την προετοιμάσει, να συζητήσουμε τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις και μετά να λάβουμε απόφαση. Όπως σας είπα όμως δεν είμαι ε, υπέρ γιατί ε, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος ε, να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε καν με αυτόν τον διάδρομο. Από πλευράς χρονικής συμμόρφωσης. Στο Ρότερνταμ Τζένοβα πάντοτε μας ελέγχθη ότι πρέπει να παρουσιαστεί σαν παράδειγμα προς μίμηση για τους διαδρόμους. Αυτή τη στιγμή όμως η Γερμανία λέει ξεχάστε το 2015, ίσως το 2021... Αυτή είναι η μία απόφαση που πήραν και τα υπόλοιπα για τους άλλους τρεις διαδρόμους δεν μπορούν να κάνουν κανένα πρόγραμμα Κανείς δεν μιλά για το πώς θα προχωρήσουν, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή και κάθε φορά που πηγαίνετε και να συστήσετε στη Γερμανία παραλαμβάνετε μία άρνηση γιατί δεν θέλουν ούτε να τα ακούσουν. Για το GSMR και το πρόβλημα των επικοινωνιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των συχνοτήτων και να διατηρήσουν ορισμένες συχνότητες για τους σιδηροδρόμους. Αλλά υποθέτω ότι αυτό που έγινε είναι ότι αυτό ήταν κάτι ενδιαφέρον για τις κυβερνήσεις και ε, οι συχνότητες είναι τέτοιες ώστε υπάρχει κίνδυνος οι προτάσεις αυτές να αργήσουν να εφαρμοστούν και να είναι εις βάρος των σιδηροδρόμων. Χρειάζεται επίσης για τις λύσεις επιπρόσθετη χρηματοδότηση, όχι εκατοντάδες εκατομμυρίων αλλά επιπλέον Λοιπόν, χρηματοδότηση η οποία μπορεί ίσως να υπάρξει και ίσως όχι. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απόφαση, το θέμα είναι σε εκκρεμότητα και Ουσιαστικά το πρόβλημα προέρχεται από τη Γερμανία. Στις άλλες χώρες έχουμε λιγότερα προβλήματα και έχουμε ήδη καλύψει τα νότα μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά το μακροπρόθεσμο όφελος του ERTMS και των διαδρόμων είναι μία αρχή που τώρα έχει γίνει αποδεκτή. Δεν αμφισβητείτε πλέον και αν θέλετε να προωθήσετε τους διαδρόμους σας πρέπει να εξετάσετε πώς είναι η υποδομή, να αφαιρέσετε τα σημεία συμφορήσεως και να έχετε μία πρώτη δημοσιογραφία ε, μια πρωτη μια λύση ε, ε, που μπορεί να γίνει γενικώς αποδεκτή. Παρακαλώ να κλείνετε γιατί τέλειωσε η ώρα σας. Εάν θέλετε λοιπόν να δείτε τι συμβαίνει, έχει γίνει μία ε, άσκηση για τον διάδρομο Α, γίνεται και για τον Γ και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μία αύξηση της ε, μεταφορικής ικανότητας 15 μέχρι 30% θα την αυξήσουμε κατά μέσον όρων 25% και συγχρόνως θα μειώσουμε και το κόστος 25%. Βάσει αυτών των προϋποθέσεων ε, μελετάμε αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε αυτό το διάδρομο. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρλο Σέκη ο οποίος είναι συντονιστής για δύο προγράμματα προτεραιότητας, το PP3 και το PP19. Και τα δύο αναφέρονται σε σιδηρόδρομο υψηλής ε, ταχύτητας. Κύριε Σέκη, έχετε και εσείς 10 λεπτά στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και επομένως θα ήθελα να αφήσω και χρόνο για τις ερωτήσεις σας. Γι' αυτό λοιπόν θα σας κάνω μια σύντομη παρατήρηση της κατάστασης έτσι όπως ισχύει σήμερα και να υπογραμμίσω επίσης και κάποιες ε, ε, συστάσεις αλλά και ε, εν τέλει κάποια συμπεράσματα τα οποία μπορώ να εξάγω για την προηγούμενη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις και για το 3 και για το 19 και θα ήθελα να υπογραμμίσω την ε, ιστορική εκκίνηση των ε, διεργασιών ε, διαλειτουργικότητας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιβηρική Χερσόνησο σε ένα τμήμα του 3. Στην πρώτη διαφάνεια λοιπόν, την οποία δυστυχώς οι ερμηνείς δεν βλέπουν, βλέπετε το ε, πρώτο κομμάτι του 3 ανάμεσα από την ε, Μαδρίτη και την ε, Βαρκελόνη που θα αρχίσει να λειτουργεί έστω με κάποια προβλήματα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την, με την περιγραφή του Μομπελιέ Νίμα. Ε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο επήγει να λυθεί. Αυτό το κομμάτι ε, του 3 θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι ε, της, του μεσογειακού διαδρόμου. Το ατλαντικό σκέλος τώρα, εδώ πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ξεκίνησε η νέα γραμμή Tour Bordeaux είναι η πιο μεγάλη εταιρική σχέση μεταξύ δημοσίου και ε, ιδιωτικού τομέα. Και πολλά θα μάθουμε από αυτή την εμπειρία, ε, η οποία επιταχύνει την εφαρμογή του ε, τμήματος του Ατλαντικού όσον αφορά την ε, Γαλλία, έστω και με κάποια προβλήματα τα οποία ακόμα πρέπει να επιληθούν όσον αφορά τη διασυνοριακή διασύνδεση Γαλλίας-Ισπανίας. Στην Ισπανία τώρα υπάρχουν αρκετές, ε, αρκετά σημαντικές ε, πρόοδοι στο βασικό κομμάτι. Εκεί το κεντρικότερο ζήτημα είναι ε, να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση στο διασυνοριακό τμήμα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τις εθνικές αρχές από την γαλλική πλευρά. Οι εθνικές αρχές προσπαθούν να το λύσουν και ευελπιστούμε ότι λύση θα εξευρεθεί τουλάχιστον στα μέσα του 12 και βεβαίως και αυτό το κομμάτι ε, θα αποτελεί τμήμα του μελλοντικού σχεδιασμού, στον μελλοντικό σχεδιασμό μάλλον θα αποτελεί τμήμα του Ατλαντικού ε, διαδρόμου. Εδώ προσπαθούμε να λύσουμε και κάποια προβλήματα διακυβέρνησης έτσι ώστε οι λύσεις να έρθουν γρήγορα. Σημαντική χρονιά λοιπόν αυτή που διανύσαμε. Το 2011 ε, σηματοδότησε σημαντικές ε, εξελίξεις. Βεβαίως του χρόνου θα έχουμε περαιτέρω βελτιώσεις ε, όσον αφορά το Ρουένσε Σαντιάγο Κορούνια, Μαδρίδ, Βαγιαδολίδ, Λιόν. Η Ισπανία λοιπόν ε, έχει προχωρήσει πολύ. Η Γαλλία προσπαθεί και αυτή να φτάσει. Ε, στην Πορτογαλία υπάρχουν κάποια ζητήματα ακόμα. είχαμε την ε, δυνατότητα ε, να ε, εξεύρουμε συνέργεια ανάμεσα στις πολιτικές και την χρηματοδότηση και επίσης με την εσωτερική των εξωτερικών του εξωτερικού κόστους επιμένουμε βεβαίως ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, υπάρχουν και ωφέλη από τη διαδικασία αυτή. Όσον αφορά τώρα το ε, κομμάτι της ε, Ιβηρικής Χερσονήσου, όσον αφορά το Priority Project 3, στην Εστρεμαδούρα είμαστε ένα βήμα πριν την λειτουργικότητα. Όμως στην Πορτογαλία βρισκόμαστε σε μια στάσιμη κατάσταση. Νομίζω, ελπίζω ότι μια λύση θα εξευρεθεί εφαρμόζοντας ε, για την ε, ώρα έναν λεγόμενο ε, διάδρομο υψηλής αποδοτικότητας, high performance, υψηλής απόδοσης, high performance corridor μέχρι τη Λισαβόνα ένας διάδρομος ο οποίος ε, θα χρησιμοποιείται εν μέρη για υψηλή ταχύτητα, εν μέρη για μεταφορά εμπορευμάτων ε, και βεβαίως ε, αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως και κατά 95% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δουλεύει πάνω στο θέμα αυτό η πορτογαλική κυβέρνηση και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί θα συμφωνία επ' αυτή της συμβιβαστικής λύσεως και ε, προσδοκούμε ότι στο μέλλον θα ευτυχίσουμε να δούμε καλύτερες λύσεις. Θα θυμάστε ίσως αυτό που είπαν οι συνάδελφοι όσον αφορά το κανάλι του Παναμά και πόσο ενδιαφέρεται η Πορτογαλία να αυξήσει τις ε, θαλάσσιες ε, μεταφορές. Βεβαίως αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μετά θα πρέπει ε, φτάνοντας στο λιμάνι κάποιος να έχει τη δυνατότητα να προωθηθεί προς τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ε, αν συνδυάσουμε το Priority Project 3 και 19 θα δείτε ότι το 19 αφορά την διαλειτουργικότητα στην Ιβυρική Χερσόνησο και εδώ βεβαίως έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες πρόοδοι όσον αφορά το κομμάτι Μαδρίτη, Βαλένσια, Αλικάντε. Βελτιώνουμε την κατάσταση όσον αφορά την, το διάδρομο της Ανταλουσίας και επίσης ε, περαιτέρω ε, πρόοδοι θα υπάρξουν του χρόνου. Ένα λεπτό ακόμα χρειάζομαι για τις συστάσεις που θα ήθελα να σας ε, υποβάλω και μετά να ακούσω τα σχόλιά σας. Όπως γνωρίζετε, στο εγγύς μέλλον το ε, μεσογειακό τμήμα θα αποτελέσει κομμάτι του μεσογειακού διαδρόμου και το αντίστοιχο θα γίνει με τον Ατλαντικό διάδρομο. Ένα μεγάλο κομμάτι έχει ήδη εφαρμοστεί και βεβαίως αυτό ε, και θα αρχίσει να λειτουργεί ο ονούπο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, λειτουργία των ευρωπαϊκών ε, διαδρόμων. Σας αναφέρθηκα και το τονίζω και το επαναλαμβάνω ότι στην Πορτογαλία έχουμε στασιμότητα και αυτό είναι πρόβλημα. Και δείξτε μου σας παρακαλώ το τελευταίο, την τελευταία διαφάνεια λέει ο, ο Βλέπετε εδώ ότι στο μέσο των Πυρηναίων υπάρχει μία διακοπή, δηλαδή ότι ε, δεν περιλαμβάνεται το τμήμα αυτό ε, στο ειδικό δίκτυο, αλλά θα αποτελέσει τμήμα του ολοκληρωμένου δικτύου. Αυτό θα γίνει αργότερα, αλλά δεν θα μετατίθεται διαρκώς, κάποια στιγμή θα γίνει. Και βεβαίως θα εξαρτηθεί και από το βάσει ποιας, στην νέα μεθοδολογία, βάσει ποιου τρόπου θα υπολογιστεί η διασύνδεση ανάμεσα στα πυρηνικά δίκτυα και τα ε, επιπλέον γενικότερα δίκτυα. Να σας πω τώρα δύο λόγια. Πέρσι στη Σαραγώσα υπεγράφει μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των τριών κυβερνήσεων, αλλά μετά δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη ε, των συμφωνιών αυτών γιατί προέκυψαν άλλα προβλήματα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ο συντονισμός και η συνεργασία είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό ζήτημα και το να προβλέπουμε λίγο το μελλοντικό ε, σύστημα των πυρηνικών δικτύων. Σας βλέπω έτοιμοι να χτυπήσετε το σφυράκι σας. Θα τελειώσω λοιπόν. Στα συμπεράσματά μου θα υπογραμμίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα προγράμματα αυτά ε, είναι λογικό λέω να υπάρχουν κάποια αμφίσιμα κομμάτια, να υπάρχουν κάποιες αμφισημίες ε, όσον αφορά ε, τα προγράμματα αυτά, γιατί είναι πολύ εμπλεκόμενοι. Γι' αυτό λοιπόν σημαντικό ρόλο παίζει η ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική. Είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας τους. Η εμπειρία μας σε μερικές περιπτώσεις μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν είχαν ξεκαθαριστεί κάποια πράγματα εξ αρχής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σέκη. Έχουμε τέσσερις ομιλητές, τον κύριο Γκρός, την κυρία Γιάλα Σάντερ, τον κύριο Τρεμόσα και τον κύριο Τρέβορ και τον κύριο Μπιλμπάου. Αλλά έχουμε μόνο τις 15 λεπτά. Και έχουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του κυρίου Σέκη. Οπότε σας παρακαλώ <clears throat> να μιλήσετε ε, για 1,5 μικρό καθένας το πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για τον συνάδελφο που θα έκανε τις ισπανικές ερωτήσεις. Εγώ θέλω να αναφερθώ εδώ μόνο εις ε, τη χρηματοδότηση διότι όπως είπατε είναι ένα από τα πιο ισχυκά προγράμματα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ό,τι δηλαδή δηλαδή επιθυμούμε όλοι. Οπότε μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ πού βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας για να είναι ένα τέτοιο ισχυρό πρόγραμμα συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Επίσης τα project bonds, τα ομόλογα ε, κατά περίπτωση ε, που αναφέρονται στα προγράμματα τα οποία επεξεργάζεστε αυτή τη στιγμή. Ε, Πώς θα μπορέσουν αυτά να βοηθήσουν την πρόθεση των προγραμμάτων και πώς διαγράφονται δεδομένα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Επίσης ανάλυση των στοιχείων κόστους παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ιδίω διότι σεβαστήκατε το χρόνο σας. Η κυρία Γιάλα Σάντερς έχει το λόγο τώρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τον κύριο Σέκη να ευχαριστήσω για όσα μας είπε και ε, όλοι αυτοί που έχουν να το κάνουν ε, ε, όσο γίνεται καλύτερα και αυτή τη διαφορά που μας έλεγαν ότι μέχρι τον Ομπελιέ μας είχαν πει όμως ότι μέχρι το 2015 θα είχε περατωθεί. Εδώ αυτά τα τμήματα στο κόκκινο κοντά στα σύνορα, ας πούμε, κοντά στην Πορτογαλία και προς τη Γαλλία, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τι γίνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι, επένδυσης, ή μήπως είναι το ότι δεν βελτιώνεται η συνεργασία ανάμεσα σε ειδικούς φορείς και στο δημόσιο, ανάμεσα στο Μπορντό, στην Ατλαντική πλευρά, ποια είναι τα προβλήματα στη Γαλλία, στους δύο διαδρόμους. Και εδώ αυτές οι ημερομηνίε που εμφανίζονται, αν είναι αξιόπιστες και τι γίνεται με αυτό το τμήμα το οποίο αναπτύσσεται το rail που είναι εναλλακτική λύση εκεί που είναι κάτι με διαφορετικούς, με διαφορετικούς διαδρόμους ε, και τι θα μπορούσε να γίνει, πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα και τη σύνδεσης με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος, ο κ. Τρεμόσα. Ναι, ο κ. Τρεμόσα. Ναι, κύριε Σέκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, την πολύ καλή σας πραγματικά εργασία. Να σας πω ότι τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής δεν θα πηγαίνουν στη Ισπανία πια. Θα υπάρξουν άλλα χρήματα για να συμπληρώσουν αυτά τα έργα και όπως ε, και προηγούμενη μελήτρια, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω για τα project bonds για αυτά τα ομόλογα έργου. Σας ευχαριστώ πάντως. Ευχαριστώ και εγώ, ο κ. Κράμερ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση και έχω σύντομες ερωτήσεις. Το EATMS είναι δικό σας πρόβλημα. Νομίζω από Ισπανική πλευρά έχουν όλα ολοκληρωθεί. Τι γίνεται με το κομμάτι της Γαλλίας και μετά νοτίως της Λιόν μέχρι τα σύνορα. Ε, έπρεπε να έχει ρυθμιστεί το 2020. Είναι δεσμευτικό. Ε, το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά μεταξύ Σαν Σεμπασιάν και Μπιλμπάου. Είναι σαφές ότι από ισπανικής πλευράς ε, αν έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι Μπορντό μέχρι σύνορα θα είναι συμβατό και βλέπω ότι κοντά στη Σαλαμάνκα υπάρχει ένα κενό. Ε, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κενό και να μην υπάρχει σύνδεση είναι γραφικό λάθος και επίσης ε, σε, αυτή, ε, την, ε, σε αυτές τις γρήγορες σιδηροδρομικές μεταφορές δεν έχει σημασία η σιδηροτροχιά γιατί η Ισπανία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο εύρος σιδηροτροχιάς που θα ισχύσει για την Πορτοκαλία. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σέκη για το σύνολο της εργασίας του και για την καλή διαχείριση όλες τις προσπάθειες που έχει αναλάβει για αυτά τα σχέδια ώστε να καταλήξουν θετικά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εδώ αυτό το διαμαρτυρικό τμήμα στα σύνορα με τη Γαλλία Μπορντό και Ντάγια και τη χώρα των Βάσκων και οι βασικές αρχές προχωρούν μέσω ενός συμφώνου διαχείρισης με τις αρχές της Ισπανίας και δεν θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση και αυτή η σύνδεση μας ανησυχεί αυτές οι δύο κόκκινες γραμμές από τα γαλλικά σύνορα και έκαναν διάφορες δηλώσεις αυτά τα τελευταία χρόνια οι γαλλικές αρχές για αυτό το έργο, για αυτό το τμήμα, για τη σύνδεση και τώρα τελευταία στον αρμόδιο υπουργό είπαν ότι θα έχουμε μια νέα αναθεώρηση, γι' αυτό πέστε μου πραγματικά ποια προβλήματα τα συναντάμε και τι γίνεται, οι τοπικές αρχές όπως εργάζονται, τι γίνεται, είναι κάτι που ατενίζει προς το μέλλον ή θα τεθεί να αμφιβόλω η αρμοδιότητα του Ισπανικού κράτους και στην περιοχή μας, στη χώρα των Βάσκων και στην Καταλωνία επίσης και εάν θεωρείτε ότι υπάρχει στο μέλλον κάποια λύση και μάλιστα συγκεκριμένα. Το θέμα της χρηματοδότησης. Υπάρχουν ήδη προβλήματα στην Πορτογαλία. Τι γίνεται, θα έχουν κανονικά μέχρι 95% ε, συμμετοχής. Αυτό συμβαίνει με την Πορτογαλία, θα μπορούσε να επεκταθεί και με άλλα τμήματα. Τι γίνεται, σας ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σέκη για να μπορέσει να μας απαντήσει. Βέβαια γνωρίζω ότι υπάρχουν λύσεις, ε, ε, ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ να είστε σύντομος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντες για τα καλά σας σχόλια. Όσον αφορά το ERTMS, η εντύπωση που έχω είναι ότι και στη Γαλλία και την Ισπανία, ιδιαίτερα δε στην Ισπανία, ε, πάει καλά και νομίζω ότι υπάρχει ικανοποίηση από αυτού. Υπάρχουν όμως ελάσσονα σημασία τεχνικά προβλήματα ε, και ο Κάρολ Βίνκ αν θέλετε μετά μπορεί να προσθέσει κάτι άλλο αφού ολοκληρώσω τα σχόλιά μου από αυτού. Για τα οικονομικά προβλήματα σε γενικές γραμμές δεν έχω τώρα χρόνο να μπω σε λεπτομέρειες, όμως ε, γνωρίζετε ότι την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη στην Αμβέρσα, θα λάβουν χώρα οι ετήσιες ε, ε, ημέρες ε, ΔΕΔ και εκεί θα γίνει ιδιαίτερο λόγος για τη χρηματοδότηση. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία και θα έχετε όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να έχετε μια επικαιροποιημένη ιδέα του τι συμβαίνει και όσον αφορά και τα ομόλογα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει. Τώρα ήδη είναι κάτι έτοιμο να ξεκινήσει. όσον αφορά το τι μπορούμε να προβλέψουμε ήδη ε, σχετικά με το Connecting Europe ε, και αυτό θα το συζητήσουμε καθώς επίσης και κάποια ε, πολιτικά και με οικονομικά στοιχεία, ας πούμε η εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους και των εξωτερικών ωφελιών βεβαίως. εσωτερήκευση λοιπόν του ωφέλους αυτό είναι πιο περίπλοκο, αλλά αδιαφυσβήτητα ε, χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, ας πούμε, το κομμάτι που θα πρέπει να υλοποιηθεί στην χώρα των Βάσκων. Ε, σήμερα υπάρχει περίπου μία ροή 10.000 βαγονιών. Εάν καταφέρουμε με τρόπο αποτελεσματικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό τότε, οπωσδήποτε να καταφέρουμε δηλαδή να μειώσουμε στο μισό τον αριθμό των βαγονιών, τότε οπωσδήποτε θα έχουμε <clears throat> μεγάλη μείωση της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Τουρ Μπορντό. καλό παράδειγμα ε, σχεδίου προτεραιότητας. Και εδώ επανέρχομαι και στο προηγούμενο σκεπτικό μου. Είναι μια καλή γραμμή γιατί είναι αποδοτική γραμμή. Επομένως η αποδοτικότητα είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό στοιχείο. Και με κάποιες ε, ε, με κάποια προσπάθεια μπορούμε να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα των προγραμμάτων. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε εντελεχέστερα στο μέλλον βεβαίως. Εγώ απλώς θέλω να σας δείξω λίγο ένα μικρό δείγμα των όσων σκέφτομαι. Όσον αφορά τώρα τον ε, μηχανισμό ε, συνοχής ε, σε σχέση με την Ισπανία λειτουργήσε πολύ καλά μέχρι τώρα και βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορθά τα υπάρχοντα χρήματα όσο τα χρήματα είναι ακόμα εδώ για την Πορτογαλία τώρα και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οτιδήποτε υπάρχει στη διάθεσή μας. Ε, να προσαρμοστούν ας πούμε οι υπάρχουσες γραμμές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες προσελήσεις οι οποίες μπορούν να είναι εποφελείς και βεβαίως ε, ε, επ' αυτού εργάζεται η Κομισιόν μαζί με την ε, κυβέρνηση της χώρας. και λαμβάνοντας βεβαίως ε, ε, υπόψη και όλες τις δεσμεύσεις που αυτή τη στιγμή έχουν υποβληθεί στα δημόσια οικονομικά της χώρας, της Πορτογαλίας. Αλλά θα ήταν πραγματικά καταστροφικό να χάσει, να χάσει μια χώρα ένα δις ευρώ ε, μια χώρα μάλιστα η οποία χρειάζεται ε, νέες επενδύσεις ε, αναζωπήρωσης της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργίας θέσεων εργασίας κτλ. για το κομμάτι της Μεσογείου υπάρχει ένα πρόβλημα με το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα και τις έγκαιρες μεταβιβάσεις, ε, κυρίως μεταξύ της Νίμ και της Λιώνα. Εκεί πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Όμως, όμως στο κομμάτι του Ατλαντικού ε, διαφαίνεται μεγαλύτερη συνένεση και έχουν αρθεί τα προσκόμματα. Είχα τη δυνατότητα τέλη Σεπτεμβρίου να ε, κάνω επισκέψεις τόπου. ξεκίνησα από τη Βρέστη. Νομίζω ότι όταν οι εθνικές και τοπικές αρχές της Γαλλίας λένε ότι δουλεύουμε ε, έτσι ώστε να εξευρεθεί ε, λύση μέχρι τα μέσα του 12 μπορούμε να τους εμπιστευτούμε γιατί όλη η διαδικασία έχει ξεκινήσει και οδηγείται προς τα εκεί. Όσον αφορά τώρα την επικοινωνία και την οικοδόμηση συνενέσεων, ναι βεβαίως όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα ερωτήματα εργαστηρίου και πρέπει σε αυτήν την έδρα να αναλυθούν. Νομίζω ότι απήντησα στις περισσότερες από τις ερωτήσεις, δεν ξέρω αν ο συνάδελφος θέλει να προσθέσει κάτι. Στην Ισπανία τα πράγματα είναι καλά, είναι σε ηγετική αν θέλετε πολύ προχωρημένη θέση όσον αφορά την ε, εισαγωγή του ε, ERTMS. Ε, δισταγμοί υπήρχαν από την πλευρά της Γαλλίας, νομίζω ότι έχει πιστεί πλέον και η Γαλλία και δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα προχωρήσει το ERTMS όπως και στις άλλες χώρες. Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους τους συντονιστές. και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον τους και τα σχόλιά τους και εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, η επόμενη θα είναι ε, συνεδρίαση θα ξεκινήσει την, ε, στις 19 Δεκεμβρίου 3 το απόγευμα ε, θα διαρκέσει δύο μέρες 20 με, 19 και 20 ακυρώθηκε η συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό μεσημέρι